Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω. Ξεκινάει η συνεδρίασή μας. Έχουμε μεταφράσει σε 23 γλώσσες, έχουμε τη μετάφραση σε 23 γλώσσες. Ταυτόχρονα οι συνεδριάσεις μας όπως ε, και σε άλλα κοινοβούλια μεταδίδονται στο διαδίκτυο και είναι ανοιχτές στο κοινό. Εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλω να σας καλωσορίσω και θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε σε αυτή την ετήσια πλέον συνάντησή μας μια συνάντηση η οποία επιτρέπει σε βουλευτές που ανήκουν στις ε, οικονομικές επιτροπές ή τις επιτροπές προϋπολογισμών κοινοβουλίων, βουλών, αντιπροσώπων και γερουσιών να συναντώνται είτε στις Βρυξέλλες είτε σε ένα κοινοβούλιο της χώρας η οποία είναι στη θέση της Προεδρίας, της εναλλασσομένης, για μια ανταλλαγή. dois vous informer du que, euh, και επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι φέτος ανταποκρίθηκαν 35 γερουσιαστές στην πρόσκλησή μας και βουλευτές που εκπροσωπούν 18 διαφορετικά εθνικά κοινοβούλια. Θα ήθελα να χαιρετήσω ιδιαίτερως τους προέδρους των Επιτροπών Προϋπολογισμών Οικονομικών από το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Ισπανία την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Φυσικά και οι υπόλοιπε χώρε εκπροσωπούνται, αλλά όχι από προέδρου κατά ανάγκη, αλλά από αντιπροέδρου ή βουλευτέ. Η σημερινή μα συνεδρίαση λαμβάνει χώρα μια ιδιαίτερη στιγμή για τη ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν από λίγες μέρες ε, είχαμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τον επόμενο Ιούνιο θα μας υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προτάσεις της για το Ευρωπαϊκό Πολιτές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μέχρι το 2020. Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια μεταβατική περίοδο και πριν από λίγες μέρες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε τη νέα διαδικασία που προβλέπει συντονισμό πολύ πιο στενό από ό,τι στο παρελθόν των 27 χωρών μελών για θέματα δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής. Και μάλιστα σε δύο-τρεις μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τις προτάσεις της για την κατανομή των βασικών τμήματων του κοινοτικού προπολογισμού μεταξύ 2014 και 2020. Το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο δηλαδή. Ξέρετε ότι ο κοινοτικός προϋπολογισμός καλύπτεται από ένα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Βρισκόμαστε στην περίοδο 2007-2013 και προετοιμάζουμε την επόμενη περίοδο των δημοσιονομικών προοπτικών 2014-2020. Γι' αυτό και θεωρήσαμε σκόπιμο και σημαντικό να διοργανώσουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων σε αυτή την κρίσιμη στιγμή του ευρωπαϊκού βίου. Γνωρίζετε ότι οι πρόεδροι των Εθνικών Κοινοβουλίων συνεδριάζουν μία φορά το χρόνο σε μια διάσκεψη κορυφή των Προέδρων των Κοινοβουλίου Και μάλιστα στην τελευταία του συνεδρίαση προσκάλεσαν και του Προέδρου ε, των Επιτροπών Προπολογισμών και Οικονομικών για συνεργασία. Και σε αυτό το πνεύμα διοργανώσαμε και τη δική μα συνάντηση. Μάλιστα σας είχαμε αποστείλει και διάφορα έγγραφα, τεκμηρίωση για την προετοιμασία αυτή της συνεδρίασης. Και αυτό που θα σας πρότεινα από μεθοδολογικής απόψεως θα ήταν μετά από, μια σύντομη, από τη σύντομη τη δική μου εισαγωγή να δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας για τον προϋπολογισμό του 2012, την κυρία Βαλτσάνη, και κατόπιν θα δώσω το λόγο στους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων που το επιθυμούν για να μας εκφράσουν τις απόψεις τους για τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης. Στη συνέχεια, και αφού ακούσουμε όλους τους εκπροσώπους που θα θέλουν να λάβουν το λόγο, σας προτείνω να συμπληρώσετε αυτό το γαλάζιο φύλλο για να δούμε πόσοι θέλουν να λάβουν το λόγο, για να μπορέσουμε να διοργανώσουμε καλύτερα την πορεία της συζήτησης και να έχουν την ευκαιρία όλοι όσοι επιθυμούν να μιλήσουν. Ως προς το υπόβαθρο τώρα της συζήτησης. Θα σας πω λίγα ενημερωτικά στοιχεία. Όλες οι χώρες βρίσκονται σε πολύ δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει προπολογισμό ο οποίος χρηματοδοτείται από τους εθνικούς προπολογισμού, εξίσου βρίσκεται σε δινήθηση. Γιατί τα χρήματα σπανίζουν όλο και περισσότερο, οπότε χρέος δικό μας είναι να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κονδύλια αυτά και να δούμε πώς, χάρη στην καλύτερη μας συνεργασία, θα υλοποιήσουμε αυτό το στόχο της αξιοποίησης ακριβώς των κονδύλιων. Πώς λοιπόν θα αποφύγουμε τις επικαλύψεις, της επαναλήψεις και άρα τη διασπάθηση των κονδυλίων, τη σπατάλη. Να αποφύγουμε λοιπόν την επικάλυψη μεταξύ των ορισμένων κοινοτικών και εθνικών δράσεων. Και σε το τομείς που πολλές χώρες αφιερώνουν εθνικά κονδύλια να χρησιμοποιηθούν καλύτερα για θέματα επιστημονικής έρευνας, για παράδειγμα. Πώς μπορούμε να συγκεντρώσουμε μια κρίσιμη μάζα, γιατί χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την επιτυχία αυτών των πολιτικών. Στόχος μας λοιπόν είναι να ξοδέψουμε λιγότερα, γιατί δεσμευόμαστε από την ε, ανάγκη εξυγίανσης και δημοσιονομικής λιτότητας, αλλά να κρατήσουμε τις απαραίτητες για το μέλλον μας δαπάνες. Πώς λοιπόν θα ξοδεύουμε καλύτερο τρόπο τα κονδυλιά μας, με μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική αποτελεσματικότητα και καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων των φορολογουμένων μας. Και επίσης πώς θα βελτιώσουμε το έργο μας και ο καθένας στην πατρίδα του, αλλά και το κοινό μας έργο, ώστε να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση των κοινών στόχων που έχουν όλες οι κοινοτικές χώρες και που συγκεντρώνονται στο πρόγραμμα Ευρώπη 2020. Το πρόγραμμα αυτό, το σχέδιο δράσης για την Ευρώπη του 2020, δεν είναι μία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μία ομόφωνη πολιτική βούληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, που υιοθέτησαν αυτή τη δήλωση τον προηγούμενο Ιούλιο. Πώς θα χρηματοδοτήσουμε λοιπόν αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το 2020. Ο κοινοτικός προϋπολογισμός συμβάλλει στην χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων αυτού του προγράμματος του 2020 και η κυρία Μπαλτσάνη θα σας παρουσιάσει το σχέδιο αυτού του μελλοντικού προϋπολογισμού αυτό που θα ήταν ενδιαφέρον είναι να μας εξηγήσει ο καθένας από εσά πώς ε, λαμβάνονται υπόψη αυτά, αυτοί οι στόχοι, αυτό το σχέδιο, αυτό το πρόγραμμα στην κάθε χώρα ή δεν λαμβάνονται υπόψη. Γιατί πριν το πρόγραμμα Ευρώπη 2020 είχαμε ένα άλλο πρόγραμμα με τίτλο «Η στρατηγική της Λισαβόνας» γιατί είχε υιοθετηθεί στη Λισαβόνα το 2000 και κάλυπτε την περίοδο 2000-2010. Ήταν μια απόφαση των αρχικών κρατών και κυβερνήσεων που όμως ε, ε, τελικά κρίθηκε ως παταγώδης αποτυχία. Αυτή τη φορά δεν έχουμε την πολυτέλεια μιας νέας αποτυχίας, γιατί τώρα μόλις βγαίνουμε από την κρίση και όχι όλες οι χώρες, μερικές ακόμη βρίσκονται εν μέσω της κρίσης, οπότε έχουμε καθήκον να εξασφαλίσουμε το μέλλον και να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα το 2020, να δούμε λοιπόν πώς θα το λάβουμε υπόψη, πώς θα το χρηματοδοτήσουμε και από το κοινοτικό υπολογισμό, αλλά και πώς τους στόχους αυτούς θα τους υλοποιήσουμε στο μέτρο του δυνατού και στην κάθε χώρα. Πώς λοιπόν μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα. Να και οι κυβερνήσεις μας στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισαν να θεσπίσουν κάποιες διαδικασίες συντονισμού των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών. Και μάλιστα έχουμε και τον όρο το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο που συνοψίζει αυτή τη διαδικασία του συντονισμού, οπότε σε κάθε χώρα η δημοσιονομική διαδικασία θα ξεκινήσει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και θα εκτιληχθεί ανάλογα με αυτά, θα αυτά που θα προβλεφθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Κάτι παράδοξο που επισήμαναν πολλά εθνικά κοινοβούλια είναι ότι μέχρι στιγμής σε αυτή τη διαδικασία που αποφάσισαν οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων δεν προβλέπεται καμία θέση για τα εθνικά κοινοβούλια. Φαίνεται θεώρησαν οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων ότι αφού ούτως ή άλλως στο τέλος του έτους τα εθνικά κοινοβούλια είναι αυτά που ψηφίζουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς, δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων από την αρχή της διαδικασίας. Πάντως η αίσθηση που ψηφιζουν τους εθνικους προυπολογισμους δεν ειναι υποχρεωτικη συμμετοχη των εθνικων κοινοβουλιων απο την αρχη της διαδικασιας παντως η αισθηση που εχουν οι περισσότεροι από εσά και την αστερνίζομαι και εγώ, είναι ότι αντίθετα θα πρέπει τα εθνικά κοινοβούλια να αναμειχθούν από την πρώτη φάση της διαδικασίας, την πρώτη μέρα της έναρξης της διαδικασίας γιατί στο Κοινοβούλιο γίνεται η δημόσια και δημοκρατική συζήτηση. Και από τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αποκτήσει και νέες εξουσίες που δεν είχε προηγουμένως και θα καθορίσει τους πολιτικούς και δημοσιονομικούς προσανατολισμούς που θα είναι κοινή πια για όλες τις χώρες, αυτές οι επιλογές θα πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο μιας πολιτικής συζήτησης σε πρώτερη φάση, πριν δηλαδή οριστικοποιηθούν αυτές οι επιλογές και στη συνέχεια θα σχολιαστούν, θα επιβεβαιωθούν ή θα απορριφθούν στις ψηφοφορίες που θα γίνουν στα εθνικά κοινοβούλια. Πολλοί από εμά πιστεύουμε ότι η διαδικασία αυτή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που αποφάσισαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είναι μια καλή διαδικασία, αλλά ανεπαρκής. Θα πρέπει να τη συμπληρώσουμε με τη συμμετοχή των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων. Και ένα από τα θέματα για τα οποία θα μπορούσαμε σήμερα το απόγευμα να συζητήσουμε είναι φυσικά η ουσία, δηλαδή πώς θα χρηματοδοτήσουμε τους μείζονες στόχους μας για το 2020, αλλά και πώς θα μπορούσαν τα Εθνικά Κοινοβούλια να αναμειχθούν ε, στη διαδικασία αυτή από την ε, πρωταρχική της φάση. Αυτά λοιπόν. Θα δώσω τώρα το λόγο στη Φραντζέσκα Μπαλτσάνη, που είναι η συγγήτριά μας, η συγγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη Επιτροπή Προϋπολογισμών για τον προπολογισμό του 2012 και θα μας παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προετοιμάζει, καταρτίζει το σχέδιο του κοινοτικού προϋπολογισμού για τα μεγάλα προγράμματα της Ευρώπης του 2020 και για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως θυμήσατε, φέτος ξεκινήσαμε τη δημοσιονομική διαδικασία για το 12 ταυτιζόμενη χρονικά με το άνοιγμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Από το 2010 είδαμε στην Ένωση πάρα πολλές χώρες να αντιμετωπίζουν δυσκολίες και ζήτησα να υπάρξουν και παρεμβάσεις για τη σταθεροποίησή τους. Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είχε δύο βασικούς στρατηγικούς στόχους. Πρώτον, να δημιουργηθεί ένα πραγματικό μέσο για μια πιο ισχυρή οικονομική διακυβέρνηση. Και επίσης να προσπαθήσουμε να πραγματώσουμε με την προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία όλες τις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε σε δημοσιονομικό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο λοιπόν από την αρχή ήταν το ε, σημείο αναφοράς θα έλεγα, ξεκινώντας ε, την προσπάθεια αυτή. Τι σημαίνει Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Σημαίνει κυρίως μία προσπάθεια για να υπάρξει μια πραγματική σύγκληση ανάμεσα στους εθνικούς προϋπολογισμούς και τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ο κοινοτικός προϋπολογισμός δεν είναι ένας απλός ε, προϋπολογισμός δαπάνης, κατανομής δαπανών μάλλον, αλλά είναι ένα στρατηγικό μέσο το οποίο επιτρέπει το συντονισμό των προϋπολογισμών των κρατών μελών. Η αντίληψη που είχαμε λοιπόν για τα δημοσιονομικά φέτος έχει γίνει η αντίληψη για μια ανανεωμένη φύση του προϋπολογισμού μας, ο οποίος θα πρέπει να είναι στην καρδιά της διακυβέρνησης και πρέπει να καταστεί στρατηγικό μέσο. Δεν είναι εύκολο να συντονίσει κανείς τον προϋπολογισμό της Ένωσης με τους εθνικούς προϋπολογισμούς, γιατί υπόκειται καταρχάς σε διαφορετικούς περιορισμούς. Υπάρχει όμως ένας ουσιαώδης συντονισμός στο επίπεδο της σύγκλησης του στόχους, της σύγκλησης στις προτεραιότητες. Σε αυτήν την προσπάθεια συντονισμού πρέπει να εμείνουμε και πρέπει να εργαστούμε και προς αυτό πρέπει να εργαστούμε. Όχι ένας τυπικός συντονισμός, αλλά ένας συντονισμός ουσίας, δηλαδή ένας στρατηγικός συντονισμός. Σήμερα οι προτεραιότητες της Ένωσης είναι ξεκάθαρες. Ε, ακολουθούμε μία στρατηγική μια στρατηγική που έχουμε προσπαθήσει σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξουμε στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020. Έχουμε σαν βασικό στόχο να εφαρμόσουμε τη στρατηγική μας αυτή σε βάθος, η οποία μέσα σε ένα αριθμό χρόνων να δώσει μετρήσιμα ωφέλη στην Ευρώπη μια στρατηγική πάνω στην οποία, πάνω στην οποία πρέπει να συγκλίνουν οι προσπάθειες με τα κράτη-μέλη. Εμείς εδώ οι πρώτοι ίσως ξεκινήσαμε την προσπάθεια να σχεδιάσουμε την κοινοτική στρατηγική, αλλά η ευθύνη όλων και των κρατών μελών είναι μεγάλη. Ο προϋπολογισμός μας λοιπόν πρέπει να καταστεί το σημείο εκκίνησης το απλό ξεκάθαρο μέσο προς το οποίο να προσβλέπει κανείς για να προσανατολίσει και τις εθνικές πολιτικές. Μην ξεχνάμε επίσης ότι το εξάμεινο το ευρωπαϊκό προβλέπει και τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα, προσπάθειες σύγκλησης δηλαδή προς το ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να εφαρμόσουμε πλήρως τις πολιτικές που αποφασίζουμε στο κοινοτικό επίπεδο. Οι στόχοι αυτοί, οι στόχοι της τραγικής του 2020 μας οδηγούν σε κάποιες σκέψεις. Πρέπει να κάνουμε μία προσπάθεια έτσι ώστε οι δημοσιονομικές πολιτικές να είναι πολιτικές μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Δεν θα πρέπει να έχουν ε, <clears throat> μία διάρκεια αυστηρά ετήσια, αλλά θα πρέπει να είναι πολιτικές στραμμένες στο μέλλον πολιτικές οι οποίες θα έχουν στόχους όχι μόνο το επόμενο δωδεκάμινο, αλλά θα προσπαθούν με αποφασιστικότητα να επιτύχουν τη σύγκληση σε μακροπρόθεσμη περίοδο. Αυτό είναι ένας επενδυτικός θα έλεγα προϋπολογισμός προς τον οποίο θα στραφεί η Ένωση. Ένας επενδυτικός προϋπολογισμός όχι μόνο γιατί οι δαπάνες της Ένωσης είναι βασικά επενδυτικές δαπάνες, αλλά γιατί το μέσο αυτό είναι θα έλεγα απαραίτητο για να συνεισφέρουμε στην προσπάθεια ξεπεράσματος της κρίσης που προκαλείται από το δημόσιο χρέος. Επενδυτικός προϋπολογισμός σημαίνει επίσης ότι θα πρέπει να είναι και η κινητήρια δύναμη των επιλογών που κάνουμε. Είναι πολύ εύκολο να το δει κανείς αντεστραμμένα όπου τα κράτη-μέλη προσπαθούν να καταλάβουν πώς είναι δυνατόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να βρουνε τους πόρους για αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν. Αντίθετα, εμείς πρέπει να κάνουμε το ανάποδο. Θα πρέπει οι πολιτικές σε εθνικό επίπεδο να καθοδηγούνται ακριβώς από τις οδηγίες τις οποίες δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πάνω σε αυτές τις οδηγίες θα βασιστούν οι χρηματοδοτήσεις που θα λειτουργήσουν σαν στρατηγικός μοχλός. Οι στόχοι της στρατηγικής του 2020 είναι η κατά στόχη του προϋπολογισμού του 2012. Αυτοί οι πέντε βασικοί στόχοι και με πρώτο στόχο έχουμε τον στόχο που αναφέρεται σε μια Ευρώπη με μεγαλύτερη και καλύτερη απασχόληση. Μια Ευρώπη η οποία να προσπαθήσει να περάσει σε μια αναπτυξιακή πλέον διάσταση. Σήμερα θα πρέπει να αναφερθούμε στη στρατηγική του 2020 σαν το μέσο που πρέπει να έχει η Ευρώπη στη διάθεσή της για να καταπολεμήσει την κρίση. Δύο είναι τα βασικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Πρώτον, να μην ξεχνάμε σε περιόδους λιτότητας και σε περιόδους δημοσιονομικής δυσπραγίας θα έλεγα, ότι η στρατηγική του 2020 δεν γεννήθηκε από το μηδέν, αλλά είναι ακριβώς απάντηση σε αυτή τη λιτότητα και είναι λύση σε αυτή την κρίση. Είναι μια στρατηγική την οποία θα πρέπει να ξεκινήσουμε να χρηματοδοτούμε άμεσα χωρίς να χάσουμε χρόνο. Γιατί η απάντηση της Ευρώπης που δίνει στην κρίση, η απάντηση που δίνει η Ευρώπη συγγνώμη, στην κρίση είναι αυτή. Έτσι θα βγούμε από την κρίση και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αρτίθεται σε κίνδυνο όπως μας ανέφερε ο πρόεδρος μας από την επιθυμία κάποιων κρατών μελών να μειώσουν τους προϋπολογισμούς επενδυτικός προϋπολογισμός που θα οδηγήσει σε μια Ευρώπη με μεγαλύτερη απασχόληση, με καλύτερη απασχόληση. Απαιτούνται επενδύσεις που αφορούν και την αγορά εργασίας αλλά και την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Μια ήπειρος η οποία αποτελείται από πάρα πολλούς νέους με προβλήματα που δεν φυσικά αφορούν μόνο τους νέους αλλά και τον υπόλοιπο πληθυσμό μια ήπειρος όπου θα πρέπει να μην φοβόμαστε τον ανταγωνισμό των αναδειωμένων χωρών. Θα πρέπει λοιπόν να επενδύουμε στην έρευνα, να επενδύουμε στην ανάπτυξη, να μεταρρυθμίσουμε με πιο σύγχρονο και δυναμικό τρόπο τις παραδοσιακές μας πολιτικές. Πολιτικές οι οποίες ήταν ένα πολύ σημαντικό βέβαια βήμα της ιστορίας μας και πρέπει να ανανεωθούν και όχι να ξεχαστούν. Είναι λοιπόν απαραίτητο να έχουμε άμεση επαφή με τους εθνικούς προϋπολογισμούς και θα πρέπει να καταστήσουμε τον κοινοτικό προϋπολογισμό ένα προσανατολιστικό προϋπολογισμό με στόχο το 2020 και να ζητήσουμε από τα κοινοβούλια των κρατών μελών να κατανοήσουν πώς είναι δυνατόν σε εθνικό επίπεδο να δημιουργήσουν τις καλύτερες συνέργειες που απαιτεί η Ευρώπη του 2020 πώς είναι δυνατόν να δράσει κανείς έτσι ώστε να υπάρξει ο απαιτούμενος ανταγωνισμός για να κλείσει ακριβώς αυτός ο κύκλος που ξεκινάει από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, περνάει από τους εθνικούς προϋπολογισμούς γιατί αλλιώς δεν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Έτσι θα δημιουργηθούν ευκαιρίες οι οποίες ξεφεύγουν από την απλή θεωρία τη δημοσιονομική και γίνονται πραγματικότητα, γίνονται ε, δικαιώματα, γίνονται πλούτος για την Ευρώπη. Merci, madame. Σας ευχαριστώ κυρία μου. Άρχισε λοιπόν η συζήτηση. Ο λόγος είναι στην διάθεση των φίλων μας εθνικών βουλευτών. Έχω δύο έγγραφα μπροστά μου. Βρισκόμαστε στο Βέλγιο. Η κυρία Βάντερ Μέρς από την Βελική Γερουσία έχει ζητήσει το λόγο. Θα δίνω το λόγο σε όποιον μου τον ζητεί. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά λαμβάνω το λόγο εδώ ενώπιον των Ευρωβουλευτών και των άλλων ε, βουλευτών για το θέμα αυτό. Πώς μπορούμε να συντονίσουμε την δημοσιονομική πολιτική. Έχει φτάσει σε κάποια όρια ο συντονισμός των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών. Ωστόσο χρειαζόμαστε περισσότερη προσπάθεια για να προωθήσουμε τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους στον σημερινό κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θεωρηθεί ως σημαντική προτεραιότητα Πρέπει να εξαντλήσουμε το οικονομικό δυναμικό που διαθέτει η Ευρώπη. Να συμβαδίσει η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς με μια ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης. Χρειαζόμαστε απλοποίηση της νομοθεσίας στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειαζόμαστε πρόσβαση σε χρηματοδότηση και υποστήριξη για τις εισαγωγές και εξαγωγές, χωρίς περιττή γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία πρέπει να μειωθεί. Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρξει αποτελεσματικότερος αγώνας κατά της οργανωμένης εγκληματικότητας. Είναι δύσκολο ωστόσο να ζητήσουμε ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες από τις ε, χώρες μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα. Η ανακατανομή των χρεών ε, με την έκδοση ευρωομολόγων αποτελεί μια δυνατότητα δεν θα πρέπει ωστόσο να οδηγήσει σε αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων και των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έπρεπε να διενεργηθεί πρώτα μια αξιολόγηση σχετικά με το κόστος από τις χώρες μέλη. Εγώ βεβαίως είμαι προσκεκλημένη εδώ, αλλά θα εκφράσω την άποψη ότι πρέπει ξανά να υπολογιστεί το κόστος για τις επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές συναλλαγές, σημαντικό και αυτό. Το Βέλγιο ενέκρινε ήδη το 2004 σχετικό νομοθέτημα τασόμενο έτσι υπέρ της φορολόγησης των οικονομικών συναλλαγών. Βέβαια, υπό την προϋπόθεση ότι και οι υπόλοιπε χώρες μέλη θα ε, ψηφίσουν σχετική νομοθεσία ή ότι θα υπάρξει ευρωπαϊκή οδηγία. Κάτι ακόμα, η οτι θα υπαρξει ευρωπαικη οδηγια κατι ακομα γυρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη εν ώψη της αυξανόμενης προσδοκίας επιβίωσης των ε, ανθρώπων στην Ευρώπη γίνεται όλο και σημαντικότερο να ε, ενισχυθεί προσπάθεια για την επιτυχία του ορίζοντα 2020 και περαιτέρω. Το ίδιο να γίνει η προσπάθεια για τον καθορισμό του ορίου συνταξιοδότησης για μας εδώ στο Βέλγιο είναι τώρα 65 ετών, βεβαίω πρέπει να υπάρξουν και κίνητρα, ώστε οι εργαζόμενοι να γίνουν και πλέον κινητικοί. Αυτό σημαίνει πάλι δυνατότητα μεταφοράς των ευρωπαϊκών συνταξιδοτικών δικαιωμάτων. Δεν θα εμβαθύνω στο θέμα αυτό αυτή τη στιγμή, αλλά χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό των εθνικών εποπτιών των χρηματιστηριακών αγορών για να μπορέσουν αυτές να αναπτυχθούν ε, βιώσιμα, γιατί και εκεί υπήρξαν πολλά προβλήματα και με την εποπτεία δηλαδή. Και εδώ χρειάζεται επομένω συντονισμό. Θα ήταν σκόπιμο να υπάρξει, για παράδειγμα, να υπάρξει και ένα δημόσιο οργανισμό αξιολόγηση τη πιστοληπτικής ικανότητα. Χρειαζόμαστε δηλαδή ένα είδο rating agency στο ευρωπαϊκό επίπεδο που να υπακούει σε ευρωπαϊκούς κανόνε το ίδιο ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο για, την, ε, για τις ε, υπηρεσίες και προϊόντα οικονομικών, ε, οικονομικού χαρακτήρα. Και αυτά βέβαια με τη συνεργασία και των φλαμανθών συναδέλφων. Σας ευχαριστώ. Όσο αφορά την τελευταία σας παρατήρηση, η θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος εποπτείας, ήδη έχουμε εξασφαλίσει αυτή την πρόταση με τρεις αρχές, μία για τις τράπεζες, μία για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και μία για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ήδη υπάρχει λοιπόν αυτός ο μηχανισμός εποπτείας. Και σε ό,τι αφορά την τελευταία σας πρόταση για έναν ευρωπαϊκό οίκο αξιολόγηση και αυτή η πρόταση συζητάται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μεταξύ των κυβερνήσεων. Θα εμβαθύνουμε περαιτέρω σε αυτή την πρόταση σίγουρα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον πρόεδρο της Επιτροπή Οικονομικών, της ε, Ισπανικής Γερουσίας στον κύριο Τζόρντι Βιλαζουάνα, γιατί αν δεν κάνω λάθος είναι καταλανικό το όνομα και άρα πρέπει να το διαβάσουμε Βιλαζουάνα και όχι Βιλαχουάνα. Πολύ σωστά κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτέ, Ευρωβουλευτέ και Γερουσιαστέ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο που μας προσκάλεσε για πρώτη φορά μετά από τη θέση εφαρμογή της Σύνθηκης Λισαβόνας για την ανταλλαγή αυτή απόψεων που είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί η οικονομική κατάσταση που ζούμε στις χώρες μας απαιτεί, όπως είπε και η συγγήτρια Μπαλτσάνη, ένα συντονισμό. Δεν έχουμε συνηθίσει σε κάτι τέτοιο, είναι κάτι πρωτοφανές και θα πρέπει να προσέξουμε και τα χρονοδιαγράμματα και το συγχρονιζόμαστε, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρη αυτή η συζήτηση και αυτό είναι το μήνυμα που θα πρέπει να διαβιβάσουμε και στις βουλές και γερουσίες μας. Εμείς συμμετέχουμε στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής για το 2020 στην Ευρώπη και μάλιστα έχουμε πολύ σημαντικούς στόχους όπως η δημιουργία θέσεων απασχόλησης που είναι ύψιστη προτεραιότητα για μας. Είναι από τις πρωταρχικές προτεραιότητες και της στρατηγικής του 2020. Λέμε ότι το 75% του πληθυσμού μεταξύ 20 και 65 ετών θα πρέπει να απασχολείται, κάτι που δεν ισχύει σήμερα γιατί έχουμε υψηλά ποσοστά ανεργίας στους νέους, μέχρι και 40% των νέων στις χώρες μας πολλές φορές είναι άνεργοι, γι' αυτό και η εξασφάλιση της απασχόλησης είναι ύψιστη προτεραιότητα και είναι πολύ σημαντικός ο συντονισμός προκειμένου να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο, ενστεριζόμαστε αυτό το στόχο για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Δεύτερο σημαντικό στόχο, να είμαστε ανταγωνιστικοί, να είναι πιο ανταγωνιστική, πιο παραγωγική και πιο αποτελεσματική η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ έχουμε δύο σημαντικού άξονε που εμφανίζονται και στη στρατηγική του 2020 και μα βρίσκουν σύμφωνου. Πρόκειται για την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη. Να είμαστε πιο ευρηματικοί, καινοτόμοι, πιο αποτελεσματική, να βελτιώσουμε την ποιότητα των προϊόντων μας και γι' αυτό χρειαζόμαστε την καινοτομία. Γι' αυτό και η ο κοινοτικό προπολογισμό έχει ως σημαντική προτεραιότητα την πρόωθηση της καινοτομία. Νομίζω ότι είναι αποφασιστικό στοιχείο αυτό για πολλούς τομείς και πολύ χρήσιμο. Κάτι άλλο που αναφέρεται στην στρατηγική του 2020 και που είναι σημαντικό είναι η κατάρτιση. Λέμε ότι δεν θα πρέπει να έχουμε ε, εγκατάλειψη της ε, φύτησης σε υψηλό ποσοστό και να εξασφαλίσουμε όσο το, όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσοστό ανώτερης εκπαίδευσης. Γιατί όσο πιο καλλιεργημένοι και μορφωμένοι είναι οι πολίτες, τόσο καλύτερη θα είναι και η κοινωνία μας. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντική προτεραιότητα, να μειωθεί η εγκατάλειψη από το σχολείο και να προωθηθεί η συμμετοχή στην ανώτερη εκπαίδευση. Επίση, θα πρέπει να συνεχίσουμε τι ε, επενδύσει στι υποδομέ, γιατί μέχρι στιγμή έχουμε επενδύσει στι υποδομέ τη Ευρώπη, έχουμε βοηθήσει χώρε να αναπτύξουν τι υποδομέ του. Βέβαια, με αποδυναμωμένου προπολογισμού ε, έχουμε πρόβλημα σε αυτό το σημείο, αλλά και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να προωθήσουμε τις επενδύσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα. Σε αυτές τις επενδύσεις να επικεντρωθούμε και να συντονιστούμε μεταξύ μας. Γιατί για την Ισπανία, για παράδειγμα, έχουμε... είναι σημαντικό το θέμα των ε, σιδηροδρομικών διαδρόμων ε, εμπορευμάτων. Ο διάδρομος τη... της Μεσογείου, για παράδειγμα. Γιατί από εκεί περνάνε το 60% των ισπανικών εξαγωγών. Είναι σημαντικός αυτός ο σιδηροδρομικός μεσογειακός διάδρομος. Και έχουμε και τον ε, Ατλαντικό διάδρομο. Για μας, λοιπόν, για την Ισπανία, η προτεραιότητα θα ήταν ε, να, συνεργαστούν και η Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προωθήσουν τέτοιου είδους επενδύσεις στις, σιδηροδρομ... στις σιδηροδρομικές γραμμές και στη μεταφορά εμπορευμάτων από τους σιδηροδρόμους. Πριν από λίγες εβδομάδες συνεδριάσαμε στην Βουδαπέστη και εκεί ακούσαμε από την Ουγγαρία την ανάγκη επενδύσεων στις ε, σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων γιατί εκεί μιλήσαμε γενικώ για την οικονομική κατάσταση και ήθεσε και η Ουγγαρία αυτή την ανάγκη να επενδύσει στις σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων. Όλοι έχουμε αρκετά στριμωγμένους ε, προϋπολογισμούς και εκεί δεν θα πρέπει να δώσουμε στον πειρασμό να περικόψουμε τις δαπάνες στις υποδομές, γιατί εκεί θα χάσουμε την ευκαιρία να κάνουμε την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο παραγωγική. Θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τις υποδομές, ιδιαίτερα τους σιδηροδρόμους, γιατί εκεί πραγματικά υπάρχει πολύ σημαντικό δυναμικό και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε με επενδύσεις. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε της Γερουσίας. Πραγματικά θέσατε το δάκτυλο επί τον τύπο των ήλων. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο. Γιατί όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε αδιανόητες για το παρελθόν εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό και σίγουρα ο μεγαλύτερος πειρασμός είναι να πλήξουμε τις επενδύσεις και θα δούμε πώς θα το αποφύγουμε αυτό, πώς θα αντισταθούμε σε αυτόν τον πειρασμό. Έχουμε το Περιφερειακό Ταμείο, έχουμε και το Ταμείο Συνοχή και αυτά τα δύο ταμεία διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Ακόμη και στη δική μου πατρίδα, τη Γαλλία, ένα τρίτο των κρατικών επενδύσεων χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Ταμείο. Και φαντάζομαι το αντίστοιχο ποσοστό σε άλλε χώρε είναι πολύ ψηλότερο στι χώρε συνοχή. Γι' αυτό και θα πρέπει να θυσιάσουμε τις επενδύσεις στη λιτότητα και να μην γίνουν οι περικοπές που θα πρέπει να κάνουμε στους προϋπολογισμούς από τις επενδύσεις μόνο. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Πάβελ Αν, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, Δημοσίων Οικονομικών της Πολωνικής Βουλής. Συγγνώμη αν κατακρεούργησα το όνομά σας. Άλλωστε η Προεδρία θα αναλάβει, η Πολωνία θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμεινο του 2011 και με την Πολωνία και την Προεδρία της θα διαπραγματευτούμε τον προϋπολογισμό του 2012. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε σήμερα μια πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα συζήτηση για το συντονισμό των δημοσιονομικών και των οικονομικών πολιτικών μας. Και θα ήθελα και εγώ να σας παρουσιάσω τις απόψεις μας. Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ως μηχανισμού διευκόλυνσης της ε, οικονομικής διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας αξιέπαινο στόχος και αξίζει υποστήριξη. Ο καλύτερος συντορισμός των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών των χωρών μελών είναι απαραίτητο ιδιαίτερα στην ε, παγκόσμια αυτή ε, δημοσιονομική και οικονομική κρίση. Θα πρέπει να περιορίσουμε τις διαφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα το σύμφωνο του ευρώ και το ευρώ συν που έχει, ε, έχει γίνει δεκτό και στην Πολωνία με ικανοποίηση. Και σίγουρα η ισχύ τη Ένωση έγκυται στην ισχυρή οικονομία τη και στο ισχυρό τη νόμισμα. Και η περαιτέρω ολοκλήρωση ε, στα πλαίσια του συμφώνου θα δημιουργήσει μεγαλύτερο δυναμικό αναπτυξιακό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα η Πολωνία θα ε, συμμετέχει ενεργά στις εργασίες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δραστηριότητες και οι εργασίες για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης και την, ε, τις πιο αυστηρές ε, διατάξεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ε, χρήζουν υποστήριξης για να αποφύγουμε μελλοντικές κρίσεις και να συμβάλλουμε στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής του 2020. Η Ευρώπη χρειάζεται να επιταχύνει την εξηγίαση των δημόσιων οικονομικών, τις μεταρρυθμίσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα και την επίσπευση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων παρόλο που η Πολωνία δεν ανήκει στην ε, Ευρωζώνη, οι διαταραχές εντός της ε, Ευρωζώνης γίνονται αισθητές και σε εμά. Γι' αυτό και οι πιο αυστηρές διατάξεις ε, και το σύμφωνο στο πλαίσιο της Ευρωζώνης και η σταθεροποίηση κατάσταση στην Ευρωζώνη είναι προς όφελος όχι μόνο της Πολωνίας αλλά και των άλλων χωρών ακόμη και δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Φυσικά θα πρέπει να ενισχύσουμε τις ε, διατάξεις της προφύλαξης στα πλαίσια του συμφώνου και να αποφύγουμε τη διόγκωση του εξωτερικού χρέους. Επίσης, ε, να εξασφαλίσουμε μια διαφάνεια των δημοσιονομικών κριτηρίων και να εξασφαλίσουμε μια συγκρισιμότητα των διαφόρων δεδομένων. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε ισότιμους όρους για την αξιολόγηση της δημοσιονομικής κατάστασης των χωρών μελών αυτών που εφάρμοσαν κάποιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και κυρίως ε, συνταξιοδοτικές. Σας ευχαριστώ. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλοι θαυμάζουμε τον τρόπο με τον οποίο η Πολωνία ήταν η μόνη από τις 27 χώρες που μπόρεσε να περάσει την παγκόσμια οικονομική κρίση χωρίς να μειωθεί το, ΕΑΠ, το εθνικό ακαθάριστο προϊόν της. Έχουμε λοιπόν πολλά να μάθουμε από το δικό σας παράδειγμα. Θα δώσω τώρα το λόγο στο Μάσιμο Καραβάλια, Καραβάλια συγγνώμη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής του Προϋπολογισμού της Ιταλικής Γερουσίας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήδη μετά από αυτά που είπε η συγγήτρια, κατανοούμε όλοι τη σημασία που έχει η καλύτερη συνεργασία ε, και ο συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών. Σε δύο επίπεδα θα πρέπει να υπάρξει αυτός ο συντονισμός. Το πρώτο επίπεδο είναι αυτό το οποίο άπτεται των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης. Το Συμβούλιο Υπουργών της χώρας μου εγκρίνει σήμερα το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων με κάποιες βασικές κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες είναι συμβατές με τις πολιτικές της Ευρώπης του 20. θα μπορούσα να βάλω σαν σύνθημα των πολιτικών αυτών είναι η ανάπτυξη χωρίς ελλείμματα. Αυτό είναι το βασικό μας θα έλεγα μέλημα. Πέντε είναι οι τομείς τους οποίους προχωράμε σε μεταρρυθμίσεις. Πρώτον προσπαθούμε να εξηγιάνουμε και να ενισχύσουμε τον προϋπολογισμό, τον κρατικό Έχουμε πετύχει αρκετά, θα έλεγα, στον τομέα αυτό, παρά τη γενικότερη κατάσταση. Το 2012 θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα έλλειμμα κάτω του 3%. Πέρυσι κλείσαμε με ένα έλλειμμα γύρω στο 4,5% από το 0, ε, κατά 0,6 κατώτερο από τις αρχικές προβλέψεις. Η δημόσια δαπάνη φέτος θα πρέπει να πέσει κάτω από το 50% σε σχέση με το ΑΕΠ. Γίνεται δηλαδή μια ουσιαστική προσπάθεια εξυγίανσης των δημοσίων δαπανών. Δεύτερος τομέας είναι η ανταγωνιστικότητα. Αύξηση της παραγωγικότητας και αύξηση της ανταγωνιστικότητας και να προσαρμοστούν οι αμοιβέ με την παραγωγικότητα. Έχουμε και άλλους τρεις τομείς παρέμβασης Αναφερθήκατε στην απασχόληση, αγορά εργασίας. Είναι μια σημαντική πρόκληση που για τη χώρα μου αφορά κυρίως τις γυναίκες και τους νέους του νότου της χώρας. Και τέλος, γίνεται μια προσπάθεια απλούστευσης για να ξεπεράσουμε θα έλεγα τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν στην αγορά και στην παραγωγή γενικότερα και στο τέλος κάνουμε μια προσπάθεια στον τομέα της καινοτομίας. Λοιπόν, αυτό το επίπεδο είναι το πιο απλό επίπεδο εφόσον θέλουμε να συντονιστούμε. Είναι το επίπεδο που αφορά την χρήση ε, των ε, ταμείων συνοχής. Σε αυτό το επίπεδο η προσπάθεια την οποία κάνει η χώρα μου αφορά από τη μία μια καλύτερη προσπάθεια συντονισμού ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένους στρατηγικούς τομείς με ε, μεγάλες, με τεράστιες υποδομές. Εδώ απαιτείται να υπάρξει μια σωστή συνεργασία ανάμεσα στα διαφορετικά θεσμικά επίπεδα. Είναι αλήθεια πως στον τομέα αυτό η συγχρηματοδότηση διευκολύνει την σύγκληση των δημοσιονομικών πολιτικών στο κράτος μέλος και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μπορεί να δημιουργεί και κάποια προβλήματα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, γιατί μπορεί να υπάρχουν πιστώσεις, αλλά δεν μπορούν να δαπανηθούν λόγω ακριβώς του Συμφώνου Σταθερότητας και προκαλούνται έτσι καθυστερήσεις στη δαπάνη. Έχει ενδιαφέρον εδώ λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προσπαθήσει να αξιολογήσει δυνατότητες πιο άμεσες, καλύτερου ελέγχου που θα επιτρέψουν από τη μία την επιτάχυνση της απορρόφησης των δαπανών, των πιστώσεων, συγγνώμη, ιδιαίτερα σε μία περίοδο που σπανίζουν οι πιστώσεις αυτές και από την άλλη να εφαρμοστεί και να ερμηνευτεί καλύτερα το σύμφωνο σταθερότητας για να αποφύγουμε αυτήν την ανάποδη επιστροφή σε σχέση με τη χρήση των φόρων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Βοσγανιάν έχει το λόγο τώρα, πρόεδρος της ε, Επιτροπής Οικονομικών της Ρουμανικής Γερουσίας. Εγώ θέλω να έρθω στον συντονισμό των εθνικών προϋπολογισμών. Βέβαια, η Ρουμανία υποστηρίζει πλήρως την στρατηγική 2020. Αυτό βέβαια δεν είναι και ε, κανένα ιδιαίτερο θαύμα, διότι όλες οι ε, χώρες υποστήριξαν την στρατηγική της Λισαβόνας, αλλά χωρίς το αποτέλεσμα που ελπίζαμε ότι θα είχε. Η γνώμη μου είναι ότι ένας από τους βασικούς ρόλους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι να γίνεται κάθε χρόνο μια αξιολόγηση για το πώς πηγαίνει η στρατηγική του 2020. Νομίζω ότι θα είναι από τους κύριους ρόλους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Εξάλλου, συζητούμε πολύ εδώ για ανταγωνιστικότητα κλπ. Η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να καθορίσουμε τον ενεργό ρόλο του προϋπολογισμού και τους μηχανισμούς που διαθέτουμε, ε, κρατικές επιχορηγήσεις, κοινοπραξίες, ε, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, μηχανισμοί κλπ. Όλα αυτά θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ε, φιλοσοφίας ενεργού ρόλου του κράτους για να προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις για σημαντικά έργα, εθνικά και ευρωπαϊκά. Για να έρθω τώρα στο θέμα όμως, η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε λίγο την εσωτερική προσέγγιση στον προϋπολογισμό. Να εφαρμόσουμε σε όλες τις εθνικές βουλές και κυβερνήσεις, να ζητήσουμε δηλαδή, να συντάσσουν ειδική έκθεση για την σύνταξη του προϋπολογισμού, ειδικά σε ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή της στρατηγικής 2020. Για παράδειγμα, η κυβέρνησή μας δημοσιεύει έκθεση για τους μακροοικονομικούς δείκτες και τη συνολική κατάσταση της οικονομίας. Θα πρέπει ωστόσο να βγαίνει και μια ειδική έκθεση για την στρατηγική 2020, την οικονομική διαχείριση κλπ. Ώστε να μας επιτρέπει να αξιολογούμε καλύτερα και να αξιολογούμε την προσέγγιση κάθε κυβέρνηση στη στρατηγική αυτή. Και δύο ακόμα πράγματα. Πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε πάνω σε μια κοινή μεθοδολογία, γιατί οι διάφοροι προπολογισμοί είναι διαφορετικοί και είναι δύσκολο να δούμε πώς θα μπορέσουν να είναι συμβατοί εφόσον οι μεθοδολογίες είναι τόσο διαφορετικές. Και μια άλλη σημαντική πτυχή. Είναι δύσκολο να υπάρξει συντονισμός μεταξύ προπολογισμών εάν κάθε χώρα ε, χρησιμοποιεί άλλο ποσοστό του ΑΕΠ. Ξεκινώντας από 32% στη χώρα μου μέχρι 48% άλλων χωρών. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο λοιπόν να τα βάλουμε όλα αυτά μαζί και να δημιουργηθεί εν τέλει μια κοινή στρατηγική και να εξευρεθούν κάποιες ομοιότητες μεταξύ της διάρθρωσης των δαπανών εφόσον τα ποσοστά του ΑΕΠ είναι τόσο διαφορετικά. Είναι δύσκολο να συγκριθούν δύο χώρες κάνουν μεταξύ τους. Μία με 32 και άλλη που έχει 45% στο ΑΕΠ. Άρα να δημιουργήσουμε όχι μόνο μια, ε, ένα, ένα κοινό σύνολο αρχών, αλλά και μια κοινή μεθοδολογία. Και τότε στο μέλλον αυτό θα επιτρέψει καλύτερο συντονισμό των προσπαθειών της κάθε χώρας για να κινητοποιήσει οικονομικούς πόρους σε σύγκριση δηλαδή με το ΕΠΤΙΣ για να επιτύχει τους κοινούς στόχους. Μάλιστα, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Λαμασούρ. Δικαίως επισημαίνεται το γεγονός ότι μέχρι τώρα το ετήσιο αυτό ραντεβού μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ε, είναι ιδιαίτερα λιτό. Ο καθένας καλείται να πει με ποιο τρόπο κάνει εξοικονομήσεις και πώς καταπίνει τέλει το πικρό χάπι. Είναι κατά κάποιο τρόπο μια ετήσια τιμωρία. Άρα δεν μπορούμε να αρκεστούμε στο να ερχόμαστε να συζητούμε πώς θα τιμωρηθούμε και απέναντι στους πολίτες μας. Πρέπει να δώσουμε και κάποια ελπίδα. Αφού λοιπόν υπάρχουν αυτά τα ραντεβού, καλά είναι να δούμε πώς κάνουμε και άλλες προσπάθειες να ζήσουμε με πιο υγιή τρόπο, να τρώμε λιγότερο για παράδειγμα και ούτω καθεξής. Να δούμε και πώς θα διατηρήσουμε την χρηματοδότηση των δαπανών στο μέλλον, ώστε για να μπορέσει να γίνει αυτό με χρήσιμο τρόπο προϋποθέτει ότι κάθε Υπουργείο Οικονομικών όταν αρχίζει να, συντάζει, να, όταν αρχίζει να συντάσει τον, το σχέδιο προϋπολογισμού να κάνει και ένα πίνακα που να επιτρέπει να δούμε ποια πράγματα από τον ετήσιο προπολογισμό χρηματοδοτούν τους μεγάλους κοινούς στόχους της στρατηγικής 2020, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στις περισσότερες χώρες αυτή τη στιγμή. Στις περισσότερες χώρες δεν έχει απολύτως καμία σχέση υπάρχει ο εθνικός προϋπολογισμός και από την άλλη μεριά ο κοινοτικός. Να πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτά μπορούν να συνδεθούν. Εάν είναι δυνατόν δηλαδή αυτό το ετήσιο ραντεβού του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα μιλήσει και για την μελλοντική χρηματοδότηση, θα πρέπει να γίνει αυτό έχοντας στη διάθεσή μας και τα δεδομένα από το εθνικό επίπεδο ο καθένας. Ε, θα βρείτε και μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον προϋπολογισμό του περσινού έτους για να δούμε ποιες, ποια κονδύλια των προϋπολογισμών χρησιμοποιήθηκαν για την ε, χρηματοδότηση των στόχων της ε, στατικής του 2020. Αυτό βεβαίως είναι για την ώρα ε, μια άσκηση επιχάρτου περισσότερο. Προχωρούμε τώρα προς τον βορρά της Ευρώπης και θα δώσω τον λόγο σε εκπρόσωπο της Σουηδικής Βουλής, τον κύριο Γιώραν Πέτερσον, της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό που είναι σημαντικό κατά με, στα πλαίσια του κοινοτικού προϋπολογισμού είναι να εξασφαλίσουμε τους πόρους για να ενισχύσουμε την ανάπτυξη στα κράτη-μέλη, γιατί όταν υπάρχει ανάπτυξη στα κράτη-μέλη, αναπτύσσεται ταυτόχρονα και ο κοινοτικό προπολογισμό, αλλά και η κοινοτική υποστήριξη ενισχύεται. Σήμερα η Σουηδική κυβέρνηση παρουσίασε στο Κοινοβούλιο του προσανατολισμού για την επόμενη διαχειριστική χρήση. Είναι ένα προπολογισμό στραμμένο προ την απασχόληση, την ε, χρηματοοικονομική σταθερότητα και την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Και αν εξετάσουμε τις μακροοικονομικές ε, πτυχές για το 2011, διαπιστώνουμε ότι θα έχουμε μία ανάπτυξη 4,6%. Θα έχουμε 0,3% πλεόνασμα και για το 2012 θα έχουμε 3 και κάτι ανάπτυξη με πλεόνασμα 3 και κάτι τεκατό. Και για το 2013 έχουμε 3,6% ανάπτυξη και πλεόνασμα 2,8%. Η οικονομική ανάπτυξη είναι αυτή στα κράτη-μέλη που θα ενισχύσει και τον κοινοτικό προϋπολογισμό και είναι μια καλή βάση για να προσεγγίσουμε τον προϋπολογισμό του 2012. Σε ό,τι αφορά τον μακροπρόθεσμο προπολογισμό τη Ένωση, στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, χρειαζόμαστε ρηξικέλευτε μεταρρυθμίσει. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη, στην οικονομική μεγέθυνση, στην καινοτομία, στην έρευνα, στην παιδεία, στην κατάρτιση και να περιορίσουμε την υποστήριξη και τις επιδοτήσεις στη γεωργία. Σε ό,τι αφορά τη φορολογία των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, η Σουηδία στη δεκαετία του 80 είχε εφαρμόσει ένα αντίστοιχο φόρο, αλλά η εμπειρία δεν ήταν καθόλου θετική. Για να λειτουργήσει ένα τέτοιο φόρο θα πρέπει να είναι παγκόσμιο και να είναι ο ίδιο για όλου. Δεν μπορεί μια χώρα μόνο ή μεμονωμένε περιοχέ να εφαρμόσουν τέτοια φορολογία γιατί με την επιβολή αυτού του φόρου οι αλλοδαπές επενδύσεις εξαφανίστηκαν από τη Σουηδία, οι επενδύσεις στράφηκαν σε άλλες χώρες και τα δημόσια έσοδα περιορίστηκαν. Ήταν πολύ αρνητική εμπειρία που είχαμε στη Σουηδία από την επιβολή του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Σε ό,τι αφορά το συντονισμό τώρα των ε, οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών, είναι πολύ καλή αυτή η πρόταση. Και στα έγγραφα που μας στείλατε, για την προετοιμασία της συνεδρίασης. Επικεντρώνομαι στα σημεία 8 και 10 και πιστεύω ότι θα πρέπει να τα αναπτύξουμε περαιτέρω και να τους δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να έχουμε ενισχυμένο συντονισμό που θα μας οδηγήσει και σε οικονομικά ωφέλη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σημειώσαμε όλα αυτά που μας είπατε και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο η Σουηδία κατάφερε για μεγάλη περίοδο να κρατήσει ψηλό ποσοστό ανάπτυξης σε σχέση με τους εταίρους της και μάλιστα μια υγιούς ανάπτυξης γιατί πολλές χώρες όπως και η δική μου πατρίδα θαυμάζουν ιδιαίτερα τις σουηδικές επιδόσεις. Και σημειώσαμε και την αρνητική εμπειρία που είχατε από το φόρο χρηματοπιστών συναλλαγών και μπορούμε να αντιλήσουμε και εμείς διάφορα διδάγματα από την σουηδική εμπειρία. Παραμένουμε στο βορρά και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του Δανέζικου Φόλκετινγκ, της Δανέζικης Βουλής, τον κύριο Όλσεν Ντύρ. Συγγνώμη πάλι που δεν προφέρω σωστά τα ονόματα. Από τη Δανική Βουλή, Φόλκετινγκ, Κυρία Όλσεν. Jeg Σας ευχαριστώ είναι σημαντικό να έχουμε συντονισμό των πολιτικών μας και αν εξετάσουμε την Ευρώπη του 2020 και τους στόχους που περιλαμβάνει, βλέπουμε ότι η σημαντική στόχη είναι η απασχόληση, για παράδειγμα. Η οικονομική μεγέθυνση, η ανάπτυξη, οι επενδύσεις στην έρευνα, στην παιδεία και βλέπουμε ότι στο σύμφωνο έχουμε περιορισμό των μισθών, περικοπές, αύξηση του, συνταξι... συντάξιμου ηλικία. Υπάρχουν ασύμβατοι στόχοι. Με τέτοιε όμω ασυμβατότητε, πώ θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε του στόχου μα, αφού είναι αντιφατικοί μεταξύ του. Κατά τη γνώμη μα, το ευρωπαϊκό εξάμεινο είναι πολύ σημαντικό. Γιατί τα θέματα του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ο εντοπισμό κάποιων μακροοικονομικών ανισορροπιών και η προσπάθεια καταπολέμησής τους είναι πολύ σημαντικό και σίγουρα χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ανάπτυξη των κοινοβουλίων. Θέλουμε περισσότερη απασχόληση στην Ευρώπη, θέλουμε ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα και εποπτεία, αλλά δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στη, στα παραδοσιακά οικονομικά μας εργαλεία και μηχανισμούς. Θα πρέπει να βλέπουμε και το γενικό πλαίσιο. Ο κοινοτικός προϋπολογισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα και τους στόχους και πρώτα απ' όλα να προσπαθήσει να υλοποιήσει τους στόχους του 2020 και θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη και λιγότερη σε παραδοσιακές πολιτικές όπως η γεωργία. Νομίζω ότι έχουμε πολύ περισσότερα να κερδίσουμε αν επικεντρωθούμε στην έρευνα και την ανάπτυξη από ό,τι στη γεωργία. Σε ό,τι αφορά το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, είναι κάτι που συζητήθηκε και στο Συμβούλιο. Ίσως ε, θα ήταν καλύτερο να εξετάσουμε μια ελάχιστη φορολογική βάση για τις βιομηχανικές και οικονομικές δραστηριότητες. Στην Δανία έχουμε πολύ υψηλό φορολογικό συντελεστή, 40% και αυτό βλάπτει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Στην Δανία εξετάζουμε αυτό το θέμα εδώ και πολλά χρόνια και δεν διαπιστώσαμε σημαντική πρόοδο. Εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει νέους πόρους, χρειάζεται και νέους ε, πόρους για να τους χρηματοδοτήσει. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον ε, Ζων Κομπέρ από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, το συμπατριώτη μου. Oui. Merci. Merci, Ευχαριστώ. Συμφωνώ μαζί, μαζί σας σε αυτό που είπατε προηγουμένως ότι ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπεται πλέον να απογοητεύσει. Μιλήσατε για την στρατηγική της Λισαβόνας. Είπατε και εσείς ο ίδιος ότι αποτέλεσε αποτυχία. Εγώ δεν θα διάλεγα ίσως αυτόν τον όρο. Αλλά ε, οι λαοί κλήθηκαν να οραματιστούν κάτι το οποίο δεν έγινε. Υπάρχει ωστόσο και τώρα μια σχετική συνένεση. Θα για την Ευρώπη του 2020 δηλαδή. Το ζήτημα είναι πώς θα φτάσουμε σε αυτήν. Και το πρώτο ερώτημα που τίθεται εν προκειμένου είναι στον βαθμό που μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές επιλογές από χώρα σε χώρα και όπου η γενικευμένη συζήτηση έγκυται στο να είπαμε ότι με την παρέμβαση των προϋπολογισμών τελικά πληρώνουν οι ίδιοι από τους συμπολίτες μας και τελικά αυτοί που έχουν περισσότερες ανάγκες. Δεύτερο, εάν για παράδειγμα γίνει με τη μείωση των υποχρεωτικών εισπράξεων, πάλι αυτό σημαίνει χρέωση. Και η χώρα μας έχει τη σχετική εμπειρία προ λίγων ετών. Άρα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυστηρή και να δούμε το θέμα των πόρων και της μεταφοράς. Γιατί στη χώρα μας είδαμε το κράτος να επιβάλλει περισσότερες ευθύνες στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Έχουμε ακόμα βέβαια πολύ δρόμο να κάνουμε για να φτάσουμε στην επιθυμητή ισορροπία αλλά έχοντα κάνει αυτή την σύντομη αυτοκριτική, θα ασκήσω κριτική και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν βλέπω τα φιλόδοξα σχέδια που ανακοινώνονται, είτε για παράδειγμα για την ε, αγροτική πολιτική, για την οποία ε, η Γαλλία τάσεται υπέρ να συνεχίσει, γιατί είναι σημαντική για την αγροτική οικονομία που είναι και από τις βασικές προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Αυτονομίας, αλλά επίσης πολιτική συνοχή, συνοχής, έρευνας, ακόμα και υποδομών. Πρόσφατα βρέθηκα εδώ σε μια συνεδρία που λοιπόν, όταν άκουσα τα φιλόδοξα σχέδια για τις υποδομές, είπα αμέσως με τον τρόπο αυτό έχουμε ξεπεράσει ήδη ολόκληρο το κοινοτικό προϋπολογισμό. Άρα χρειαζόμαστε κάποιο βαθμό συντονισμού να μην θεωρούμε ότι μπορούμε να ανακοινώνουμε φιλόδοξα, σχέδια και θεωρώντας ότι θα πληρώσουν οι άλλοι. Με τα λόγια μου αυτά απευθύνω έκκληση και για να αποφύγουμε νέα χρέωση. Βλέπε, εκτός εάν τα ευρωμόλογα είναι πραγματικά, είμαστε βέβαιοι ότι είναι μια επένδυση για το μέλλον διότι αν δούμε όλες τις επενδύσεις στο μέλλον του παρελθόντος, ίσως θα εκπλαγούμε πολύ οδυνηρά. Σας ευχαριστώ κύριε συνάδελφε και συμπατριώτη. Πράγματι, οι μελλοντικέ επενδύσεις του παρελθόντος μας έχουν προλάβει. Είναι ζήτημα φιλοσοφικό. Είναι βέβαια προφανές ότι η σωστή χρήση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και με την υποβολή αριθμητικών στοιχείων. Πήρατε ένα καλό παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την συνήθεια να λέει ότι για την διασφάλιση της υλοποίησης του συνόλου των ε, μεταφορών προσώπων και εμπορευμάτων και ενέργειας και τηλεπικοινωνιών είναι της τάξης των 200 300 δις ευρώ για τα επόμενα δεκαέτια. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα όμως, διότι συγχαίουμε χρηματοδοτήσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, για παράδειγμα για τους αυτοκινητοδρόμους, εξ αντιθέτου υπάρχουν τομείς όπου είναι απαραίτητο να χρηματοδοτηθούν από τα δημόσια ταμεία για να υπάρξει πρόοδος. Βέβαια, θα γίνει πολιτική συζήτηση μόνο εφόσον τα πράγματα είναι απόλυτα ξεκάθαρα όπως επιμείνατε και εσείς να τονίσετε. Ο κύριος Νέγκρι από το Λουξεμβουργικό Κοινοβούλιο. Επιτροπή Οικονομικών. Ευχαριστώ. Είναι σημαντικό να ενισχύσουμε τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη. Αλλά ας μην ξεχνούμε και το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Μετά το πυρηνικό ατύχημα της Ιαπωνίας, μήπως θα πρέπει να προσανατολίσουμε διαφορετικά την ενεργειακή μας πολιτική. Στο παράρτημα 5 βλέπουμε 43,7% για κλείσιμο εργοστασίων από την ατομική υπηρεσία. Και μήπως έτσι όμως θα περικοπεί ο προϋπολογισμός για το ΙΤΕ, για τον πειραματικό θερμοπυρηνικό αντιδραστήρα. Ίσως ο προϋπολογισμός μας μέχρι το 2020 θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο σε θέματα έρευνας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προκειμένου να βρούμε μια καλύτερη ισορροπία ενεργειακή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε αγαπητέ συνάδελφε. Όντως είναι ένα θέμα που θα μας προβληματίσει στα πλαίσια των στόχων του 2020. Ολοκληρώνουμε λοιπόν αυτό το γύρο των εκπροσώπων των Εθνικών Κοινοβουλίων με την κυρία Γκέρκενς που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βελγικής Βουλής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εστερνιστώ καταρχήν τη δική σας ανησυχία σε ό,τι αφορά την ανάμειξη των Εθνικών Κοινοβουλίων σε πρόορη φάση της διαδικασίας, ιδιαίτερα της ε, διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Γιατί αν ο τρόπος που μια χώρα υλοποιήσει τους στόχους και οργανώσει τον προϋπολογισμό της προσκρούσης σε αντιρρήσεις του Συμβουλίου, θα πρέπει να διορθωθεί αυτός ο εθνικός προϋπολογισμός. Ένας προϋπολογισμός όμως που καταρχήν θα έχει εγκριθεί από την αντίστοιχη Βουλή. Γι' αυτό και είναι σκόπιμο να ενταχθεί, ενταχθούν τα εθνικά κοινοβούλια σε προγενέστερη φάση της διαδικασίας γιατί μέχρι στιγμής δεν είναι προφανές πώς θα καταφέρουμε εμείς να προσανατολίσουμε τις εθνικές πολιτικές με βάση τις, το feedback που θα έχουμε από το ευρωπαϊκό επίπεδο, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις στο Συμβούλιο. Αυτό πραγματικά είναι κάτι που μας ανησυχεί ιδιαίτερος και είναι ένα θέμα που το εξετάζουμε με με την κυβέρνησή μας, παρόλο που το θέμα της βελγικής κυβέρνησης βέβαια είναι ένα άλλο φλέγον ζήτημα αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να εξετάσουμε και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να καθοδηγήσει και να υποστηρίξει τις εθνικές πολιτικές για να υλοποιήσουν τους στόχους της στρατηγικής του 2020. Είναι προφανές ότι είναι αναγκαίος ένας επαναπροσανατολισμός των οικονομιών μας και ως προς τον τρόπο παραγωγής αλλά και ως προς το είδος των προϊόντων που θα μας εξασφαλίσουν μια πιο βιώσιμη και φιλοπεριβαλλοντική ανάπτυξη, πιο οικολογική. Αλλά καλό θα ήταν και πιο ενδιαφέρον να αναβαθμίσουμε και τον κοινοτικό προπολογισμό για να μπορέσει πραγματικά να οθήσει και τις εθνικές οικονομίες προς επενδύσεις που θα προωθήσουν την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά θα ενισχυθούν και οι διασυνοριακές επενδύσεις, γιατί έχουμε τα δίκτυα μεταφορών και τα ενεργειακά δίκτυα, αλλά έχουμε και τους κλάδους της ενεργειακής αποδοτικότητας, των ανανεώσιμων ποιών ενέργειας και αυτοί οι τομείς χρήζουν επενδύσεων. Υπάρχει και το θέμα επίσης της περιφερειακής πολιτικής. Αν στο Βέλγιο δεν έχουμε αυτή την ευρωπαϊκή βοήθεια και τους ευρωπαϊκούς προσανατολισμούς, ακόμη και αν αισθενιζόμαστε αυτούς τους στόχους και έχουν αντίκρισμα στις πολιτικές μας, θα είναι δύσκολο να τους υλοποιήσουμε αν δεν υπάρχει μια γενικότερη πανευρωπαϊκή πολιτική και κάλυψη. Έτσι θα, θα υλοποιήσουμε πιο εύκολα τους στόχους μας, γιατί οι οικονομίες κλίμακος απαιτούν πιο σημαντικούς πόρους, αλλά και συνεργασία μεταξύ των γειτονικών χωρών. Αυτό που μας, που μας ανησυχεί αυτή τη στιγμή και στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, αλλά και στις συστάσεις οικονομικής διακυβέρνησης, αλλά και με το Σύμφωνο για το Ευρώ, είναι ότι η θέση των κρατικών επενδύσεων και στην έρευνα, στην καινοτομία, στην παιδεία, στην υγεία και στην καταπολέμηση της φτώχειας, γιατί και αυτή είναι στόχη της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το 2020, αυτές οι δημόσιες δαπάνες θεωρούνται ως επενδύσεις και όχι ως κρατικές δαπάνες που βαρύνουν τον προϋπολογισμό. Οπότε είναι λογικό να υπάρχει μια διαφάνεια και σε αυτή την περίοδο λιτότητας και οικονομιών που απαιτούνται θα πρέπει παρόλα αυτά να έχουμε και πιο μακροπρόθεσμες επενδύσεις που θα φανεί η απόδοσή τους και το όφελός τους μερικά χρόνια αργότερα. Εκεί μερικές φορές έχουμε ανησυχίες γιατί ακούμε για την ανάγκη μισθολογικής ανταγωνιστικότητας, ε, συνταξιοδοτικής ανταγωνιστικότητας, ε, ε, επενδυτική ανταγωνιστικότητα και ταυτόχρονα περικοπών των δημοσίων οικονομικών και περικοπής των προϋπολογισμών που αναφέρονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει μια μικρή συμβατότητα, γι' αυτό και είναι σημαντικό να έχουμε συντονισμένες πολιτικές και συνεπείς πολιτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί μόνο έτσι θα καταφέρουμε να εξηγήσουμε αξιόπιστα στους πολίτες ποιοι είναι οι στόχοι μας. Και δεν θα πρέπει απλώς να εμένουμε σε αρχές της ε, απελευθέρωσης ε, των, ε, ή των δημοσίων επενδύσεων και σε γενικά λόγια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλες οι εθνικές βουλές που εκπροσωπούνται έχουν ήδη λάβει τον λόγο. Έχω και άλλε αιτήσει λήψης λόγου από εθνικούς βουλευτέ, αλλά ας περάσουμε τώρα στους ευρωβουλευτέ. Κοντά μας είναι η κυρία Μπερέ, που στα πλαίσια της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής είναι η συγγήτρια για την διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αντίθετα από άλλε εθνικέ βουλέ, έχουμε δύο αρμόδιε επιτροπέ, την Επιτροπή Προπολογισμών και την Οικονομική και Νομισματική. Η ε, κυρία Μπερέ ε, έχει πολλέ ιδιότητε. Ε, είναι και πρόεδρο τη Κοινωνική Επιτροπή. <clears throat> Και βεβαίω, όπω σα είπα πριν, ασχολείται με το θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά βέβαια τις αρμοδιότητες των εθνικών βουλών, εδώ έχουμε ίσως μια ε, δυσυπόστατη ε, προσέγγιση. Εσείς έχετε τον προπολογισμό, αλλά η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή εξετάζει τους προϋπολογισμούς των, ε, των χωρών μελών και ιδίως την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Στα πλαίσια της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής όντως ανέλαβα την εισήγηση αυτή ιδίας πρωτοβουλίας όπως ε, αποκαλείται για την πρωτοβουλία αυτή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Δεν πρόκειται επομένω για ουσιώδη έκθεση για την ώρα, αλλά για το ερώτημα πώς είναι δυνατό με αυτή την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσπαθήσουμε να πλαισιώσουμε μια συζήτηση δημοσιονομικού χαρακτήρα των χωρών μελών στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Να εξετάσουμε πώς μπορούμε δηλαδή να συνεργαστούμε. Έχουν αναλυθεί ορισμένες πρωτοβουλίες είτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε στις Εθνικές Βουλές για να υπάρξει μια πολιτική έκφραση, έκφραση πολιτικής βούληση κάποια στιγμή. Όταν εξετάζω το χρονοδιάγραμμα, όπως φαίνεται να διαγράφεται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι αρχές του έτους, τον Ιανουάριο δηλαδή, θα καταθέσει ένα έγγραφο αναφοράς που θα είναι η ετήσια έκθεση ε, ανάπτυξης. Θα είναι τώρα όμω αυτό έγγραφο περισσότερο το οποίο θα εξετάσει το τι έχει συμβεί, δηλαδή το προηγούμενο έτος, ή θα είναι μάλλον κάτι το οποίο θα δίνει τους προσανατολισμούς για το ερχόμενο έτος. Το δικό μου προέστημα είναι ότι μάλλον θα είναι και τα δύο. Πάντως είναι κάτι το οποίο ε, πρέπει να συζητήσουμε και με εσά αλλά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην βάση του εγγράφου αυτού, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή Αρχηγή Κρατών και Κυβερνήσεων, στη διάρκεια του Εαρινού Συμβουλίου, τον Μάρτιο δηλαδή, θα εγκρίνουν ένα πλαίσιο αναφοράς των ε, προϋπολογισμών των χωρών μελών, οι οποίοι προϋπολογισμοί των χωρών μελών θα προκαθοριστούν από τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων που αυτή τη στιγμή εκπονούνται στις χώρες μέλη και βεβαίως η ικανότητα παρέμβασης που έχετε πριν να καταθέσουν τα προγράμματα αυτά οι χώρες μέλη θα είναι περιορισμένη. Δεν θα πω βεβαίως στις δικές σας διαδικασίες, αλλά κατανοώ ότι υπάρχει και αυτή η διάσταση που σας ε, ανησυχεί. Ε, εδώ τώρα στην Επιτροπή Προϋπολογισμών της Ευρωβουλής Υπάρχει μια διάσταση που ε, μας απασχολεί πολύ και όπου χρειάζεται να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Πώς δηλαδή αυτή τη στιγμή θα έχουμε συμφωνήσει επί της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι προϋπολογισμοί των χωρών μελών θα μας επιτρέψουν να είμαστε συμπληρωματική στρατηγική αυτή, γιατί ο κοινοτικός προπολογισμό δεν είναι επαρκής ώστε να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για να κινητοποιήσει ολόκληρη αυτή τη στρατηγική. Παράδειγμα, το θέμα της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ανάπτυξης. Γνωρίζουμε ότι αν θέλουμε να κερδίσουμε την μάχη των επόμενων ετών, το θέμα αυτό είναι σημαντικό, απόλυτα σημαντικό. Στη συζήτηση <clears throat> του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν κονδύλια όπου αυτά μάλλον θα είναι κονδύλια όπου θα πρέπει να τους αποδώσουμε ε, ιδιαίτερη σημασία. Αν όμω οι προπολισμοί των χωρών μελών κινηθούν σε μια τελείως διαφορετική στρατηγική, αυτό βεβαίως προκαλεί σημαντικές δυσχέρειες. Η κρίση που περνούμε τώρα και οι πρωτοβουλίε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με αυτό το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο μας υποχρεώνουν να βρούμε και τον πολιτικό χώρο για να συζητήσουμε, να διεξάγουμε δημόσια συζήτηση των μεγάλων ε, πολιτικών και οικονομικών προσανατολισμών, αλλά και να σκεφτούμε επίσης πώς θα εξασφαλίσουμε μια συμπληρωματικότητα μεταξύ του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των χωρών μελών. Εξού και η πρόταση παρέμβασης και η πρόσκληση μάλλον να παρέμβω στην συζήτησή σας, για την οποία ευχαριστώ τον Πρόεδρο που με έδωσε το λόγο τελικό, τελευταίο μάλλον σχόλιο. Βλέπω ότι σήμερα στο πνεύμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θίγει μόνο τυπικά μια κοινοβουλευτική διάσταση. Εγώ, εγώ θεωρώ ωστόσο ότι εναπόκειται στις Εθνικές Βουλές και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να καθορίσουν τα ίδια την θέση που θα έχουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Η διαδικασία αυτή δεν είναι απλώς μια διαδικασία η οποία θα οδηγήσει σε γραφειοκρατικές ε, κυρώσεις, αλλά είναι ένα πολύ πολιτικό πλαίσιο, ένας χώρος πολιτικός όπου θα συζητηθούν οι δημοσιονομικές πολιτικές. Αν αυτές λοιπόν δεν συζητηθούν δημόσια μέσα στα πλαίσια μια συζήτηση με πολιτικό χαρακτήρα, φοβούμε ότι υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι και για την λειτουργία των δημοκρατιών μας. Αυτές είναι λίγες σκέψεις που επιθυμούσα να εκφράσω και με αυτές να παρέμβω στη σημερινή σας συζήτηση. Ευχαριστούμε, Περβάς. Tout le monde a bien compris qu'avec cette de ce... Με αυτή τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σπίστηκε ένας τελείως καινούριος μηχανισμός. Τα σχέδια ή τα προσχέδια των εθνικών προϋπολογισμών θα υποβάλλονται πια σε συζήτηση και σε ανάλυση, εξέταση και κρίση στις Βρυξέλλες. Προσοχή όμως. Θα γίνεται συζήτηση στις Βρυξέλλες, αλλά όχι από τις Βρυξέλλες. Δηλαδή, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κρίνουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Η κάθε χώρα θα κρίνει τους προϋπολογισμούς των υπόλοιπων χωρών. 27 υπουργοί ΕΚΟΦΗΝ και 27 πρωθυπουργοί θα συνεδριάσουν για να εξετάσουν και να κρίνουν από εκείνο τους προϋπολογισμούς τους. Η Επιτροπή θα δώσει μια γνώμη. Αλλά δεν είναι τα κυρωτικά θεσμικά όργανα που θα λάβουν την απόφαση. Αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι. Δεν είναι κοινοτική η μέθοδος. Είναι μια κοινή εξέταση των εθνικών σχεδίων προϋπολογισμών. Αλλά, υπάρχει ένα αλλά όπως είπατε και πολύ, εκεί που ανακύπτει το πολιτικό πρόβλημα είναι ότι αν δεν υπάρξει επίσημη παρέμβαση των κοινοβουλίων, ιδιαίτερα των εθνικών κοινοβουλίων, δεν θα έχουμε δημόσια συζήτηση. Και οι προσανατολισμοί του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ δεν θα έχουν γίνει κατόπιν δημόσια συζήτησης ή ψηφοφορίας, έστω και ενδεικτικής, σε μια Βουλή. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα δημοκρατικής νομιμοποίησης και εύρεθμης λειτουργίας που οδηγούν στη λήψη αποφάσεων που βρίσκονται στο επίκεντρο των κρατικών πολιτικών. Και εκεί είναι που θα πρέπει να εξετάσουμε και να προτείνουμε ένα τρόπο διόρθωσης αυτής της ανισορροπίας και κάλυψε αυτού του κενού, ώστε το συντομότερο δυνατό και σε αρχική φάση να εντάξουμε και μία κοινοβουλευτική συζήτηση, μία ανοιχτή δημόσια συζήτηση με τη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Οι υπηρεσίε Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν εκπονήσει ένα έγγραφο που περιγράφει σε ένα πίνακα, ένα χρονικό πίνακα από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο παρουσιάζει τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και δεν φαίνονται πουθενά τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτό πραγματικά είναι αδιανόητο και απαράδεκτο. Ξεκινάμε με μια ετήσια έρευνα της Επιτροπής για την Ανάπτυξη. Μετά έχουμε την ε, συζήτηση προσανατολισμού στο Συμβούλιο Υπουργών, στο ΕΚΟΦΗΝ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα γίνει συζήτηση. Ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέχεια συζητάμε άλλωστε. Αλλά δεν είναι ο δικό μα προπολογισμό εδώ που θα εξετάσουμε, είναι οι δικοί σα προπολογισμοί που θα εξεταστούν στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ. Μετά ε, το Μάρτιο θα έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τη διάσκεψη κορυφή και στα μέσα Απριλίου σε κάθε χώρα θα υιοθετηθούν τα εθνικά προγράμματα σταθερότητα και σύγκληση. Εκεί φαντάζομαι ότι, ξέρατε βέβαια από κάθε χώρα, αλλά εκεί φαντάζομαι ότι θα έχουν κάποιο λόγο τα εθνικά κοινοβούλια στην υιοθέτηση των ε, προγραμμάτων. Αλλά βρισκόμαστε ήδη στα μέσα Απριλίου και αυτή η συζήτηση στα κοινοβούλια θα ακολουθήσει τη συζήτηση της διάσκεψης κορυφής. Υπάρχει πρόβλημα εδώ που μπορεί να είναι και πολύ σοβαρό. Γιατί βλέπουμε ότι αν δεν γίνει εκτενής δημόσια συζήτηση στα κοινοβούλια μας για τις σημαντικές αυτές επιλογές που γίνονται εγκρυπτό και παραβίστο και κλεισμένο το θυρών από τους ηγέτες μας, κάποια στιγμή θα εξεγερθούν οι, πολίτες ή η κοινή γνώμη. Και αν οι αποφάσεις ήταν δημοφιλείς ή ευχάριστες γενναιόδορες, ε, γίνεται κατανομή του πλούτου με αιτήσια ποσοστά ανάπτυξη 10%, πολύ ωραία. Αλλά δυστυχώς δεν θα είναι αυτή η κατάσταση τόσο ρόδινη τα επόμενα χρόνια, δεν θα είναι ευχάριστες αυτές οι επιλογές. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να επέμβουμε. Ήδη από την πρώτη μέρα, αν είναι δυνατόν, με ανάμειξη και των Εθνικών Κοινοβουλίων σε όλη την πορεία της διαδικασίας, προκειμένου να εξασφαλίσουμε μια διαφάνεια και μια δημόσια συζήτηση από την αρχή με ρόλο όλων των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και άλλοι έχουν ζητήσει το μεταξύ το λόγο και από την Εθνικά Κοινοβούλια. Φυσικά και οι Ευρωβουλευτές έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν γιατί είμαστε όλοι ίσοι εδώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Νίτο Αντριάν από τη Ρουμανική Βουλή. Ο κύριος Αντριάν είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι έχω υπεράσει περίπου το μισό ευρωπαϊκό εξάμεινο και μιλάμε για την διακοινοβουλευτική συνεργασία στον τομέα των δημοσιονομικών. Στην πρόσφατη συζήτηση που έγινε στο κοινοβούλιο σας επίσης Υπάρχει μία θα έλεγα θεσμική ζήλια, ένας θεσμικός φθόνος ανάμεσα στα κοινοβούλια debate has all condition to be efficient and to bring its contribution to European economic governance. Υπάρχει εκεί ένας διαφορετικός τρόπος που βλέπει ο καθένας τον ρόλο των κοινοβουλίων των κρατών μελών και <clears throat> δεν υπήρξε συγκεκριμένη αναφορά στο ρόλο των κοινοβουλίων. Όπως είπε ο Ιταλός συνάδελφος νωρίτερα, οι στόχοι της στρατηγικής του 2020 στην ουσία απορροφούν τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα, όπως και τα προγράμματα σταθεροποίησης και τα προγράμματα συνοχής, τα οποία πρέπει να παρουσιαστούν και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2011 τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να λειτουργήσουν, θα έλεγα, με συγκλίνοντα τρόπο και συμπληρωματικά. Γιατί μέχρι τώρα ε, υπήρχε μια απόκληση μεταξύ τους και στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις. Στη Ρουμανία η κυβέρνησή μου πρέπει να παρουσιάσει τη δημοσιονομική της στρατηγική για το 2012-2014 στη Βουλή. θα γίνει προσπάθεια να επηράσει ένας νόμος ευθύνη όπως λέγεται στη χώρα μου για τα δημοσιονομικά και η συζήτηση θα γίνει και σε αυτή τη φάση στη Ρωμανική Βουλή. Η στρατηγική αυτή θα εγκρίνει τα μέσα ανώτατα όρια, τα ανώτατα όρια μάλλον για ορισμένες πολιτικές και στον τομέα του, του δημοσίου χρέους και στον τομέα των ελλημάτων. Θυμίζω επίσης ότι έχουμε στη Ρουμανία και ένα εθνικό ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο, το οποίο προτείνει την υποστήριξη των κυβερνητικών προτάσεων και τεκμηριώνει τις προτάσεις αυτές, προωθώντας ταυτόχρονα την διαφάνεια στον τομέα των δημοσιονομικών. Η δημοσιονομική στρατηγική μαζί με τον νόμο για τον καθορισμό των δικτών για το 2012 θα γίνει αντικείμενο συζήτηση στα τέλη Μαΐου αρχές Ιουνίου. Με αυτή την αφορμή μπορούμε να ελέγξουμε κατά πόσον οι στόχοι της Ευρώπης του 2020 αντικατοπτρίζονται στις ε, διατάξεις του προϋπολογισμού όπως θα ε, το ζητάει επίσης το ίδιο και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Στο εσωτερικό της Ευρωζώνης η κοινοβουλευτική συμμετοχή μερικές φορές περιορίζεται σε μια ε, προσανατολιστική συζήτηση την άνοιξη. Αλλά παρόλα αυτά Υπάρχουν συζητήσεις σε διάφορα επίπεδα για τα προγράμματα σταθεροποίησης όπως επίσης ε, ε, και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οποία θα καταθέσουμε προτάσεις και συστάσεις. Ο ρόλος των κοινοβουλίων παραμένει λοιπόν και στα πλαίσια του πρώτου εξαμήνου, του πρώτου ευρωπαϊκού εξαμήνου. Η πρότασή μου είναι να εμπλακούν ακόμα περισσότερο τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια ήδη από το μήνα Φεβρουάριο ιδιαίτερα στα πλαίσια των εθνικών προγραμμάτων σύγκλησης. Η συζήτηση αυτή, αυτή είναι η πρόταση που κάνουμε για τη χώρα μου βέβαια, γιατί κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανόνες αλλά η ανάλυση των τομεακών πολιτικών στα πλαίσια το, του εσωτερικού των προγραμμάτων αυτών θα γίνει από τις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου της χώρας μου. Τι άλλο να σας πω. Πράγματι είναι μια καλή πρόταση σε σχέση με το τι συμβαίνει κυρίως στη χώρα σας, θα το λάβουμε υπόψη. Πάμε τώρα στη Σουηδία. Σφενέρικ Μπούκτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Λέγομαι Μπούκτ. Είμαι μέλος της Επιτροπής ε, Οικονομικών, όπως και ο προηγούμενος συνάδελφος. Η σουηδική θέση σε σχέση με τον προϋπολογισμό σε κοινοτικό επίπεδο είναι πολύ γνωστή έχουμε μια περιοριστική θα έλεγα αντίληψη σχετικά με το ρόλο του κοινοτικού προϋπολογισμού. Έχουμε ίσως λόγους για να το κάνουμε αυτό. Γιατί το λέμε αυτό. Περνάμε δύσκολες περιόδους στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν δημοσιονομικές περικοπές, δραστικές σε ορισμένες χώρες και στα δημόσια οικονομικά και αυτό είναι κάτι που θίγει τον ευρωπαϊκό πληθυσμό ο οποίος καλείται να χρηματοδοτήσει τα συστήματα όπως της κοινωνικής ασφάλισης. Όταν μειώνεται λοιπόν η κάλυψη κοινωνική ή όταν χάνονται θέσεις απασχόλησης, τα πράγματα χειροτερεύουν. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κρίσιμη φάση. Και είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρχουν αντιδράσεις και στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο βέβαια. Βιώνουμε μια δραματική χρονιά. Διαδηλώνουν οι πληθυσμοί σε όλες τις χώρες, στον τρίτο κόσμο και στην Ευρώπη. Χιλιάδες ε, διαδηλωτές είναι στους δρόμους και διαμαρτύρονται. Η προσπάθεια την οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συγκεντρώσει την προσοχή της και πρέπει να στοχεύει τον Ευρωπαίο πολίτη. Θα πρέπει να συντονιστούμε ακόμα περισσότερο λοιπόν. Ο συντονισμός είναι μια καλή πρόταση. Ταυτόχρονα θα πρέπει να καταστήσουμε την δραστηριότητά μας πιο αποτελεσματική. Θα πρέπει να επιταχύνουμε τη δραστηριότητά μας σε ορισμένους τομείς και να την επιβραδύνουμε σε άλλους. Την απασχόληση πρέπει να επιταχύνουμε και πρέπει να επιβραδύνουμε σε κάποιους άλλους τομείς όπως στην Γεωργία και να μεταφέρουμε τις διαθέσιμες πιστώσεις προς τη δημιουργία των θέσεων απασχόλησης. Δεν θα πρέπει οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες. Η καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων δεν θα πρέπει να χωρίζεται στα δύο ανάμεσα σε αυτούς που εργάζονται και σε αυτούς που βρίσκονται στην ανεργία. Η απασχόληση είναι η βασική μας προτεραιότητα ανεξάρτητα από τη δημοσιονομική κατάσταση. Η κακή δημοσιονομική κατάσταση δεν είναι άλοθη ε, για να μην δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Μέσω της κατάρτισης φυσικά, μέσω της εκπαίδευσης και μέσω της επένδυσης στις νέες ε, τεχνολογίες και στις ε, διεθνείς και ευρωπαϊκές υποδομές οφείλουμε να λειτουργήσουμε δίδοντας κίνητρα έτσι ώστε τα εθνικά δημοσιονομικά να γίνονται αντικείμενο προσεκτικής ε, στήριξης και φυσικά θα πρέπει να υπάρξει απαιτούμενη συνδρομή όπου χρειάζεται για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Στόχος είναι να δημιουργηθούν ορισμένες νομικές ρυθμίσεις οι οποίες θα επιτρέψουν να ελέγξουμε και κάπως καλύτερα τις, ε, τα χρηματοπιστωτικά γενικά και τα τραπεζικά προβλήματα τα οποία ε, μας κόστησαν πάρα πολύ και ο Ευρωπαίος πολίτης δεν θέλει να ξαναπληρώσει γι' αυτά. Θα πρέπει να υπάρξει επίσης και σωστή κατανομή των ευθυνών σε διεθνές επίπεδο, στον τομέα της αγοράς εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης, της φορολογίας, Αυτά όλα δεν ξέρω αν θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο αντιμετώπιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να είναι ομοσπονδία. Είναι ένα σχέδιο γενικότερα συνεργασίας. Θα πρέπει στα πλαίσια αυτού του σχεδίου συνεργασίας να μην δημιουργούνται προβλήματα και να μην προκαλείται η δυσαρέσκεια των Ευρωπαίων. Πρέπει να εμείνουμε στην πολιτική για την απασχόληση πάντως. Ευχαριστώ συνάδελφε. Σούριαν από την ε, Ουγγαρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο σύντομες παρατηρήσεις, παρακαλώ αν με επιτρέπετε, σε σχέση με, τις, με τα όσα ανέπτυξαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Βέβαια, μου αρέσει, χαίρομαι πολύ που μπορώ και συμμετέχω στην παρούσα συνάντηση δεν είναι κάτι που μας επιβάλλατε. Πραγματικά έχει νόημα η συνάντηση αυτή. Η πρώτη μου παρατήρηση αναφέρεται στην πρόταση να δοθούν περισσότερα χρήματα για την ε, έρευνα και καινοτομία. Εγώ συμφωνώ απολύτως. Θεωρώ ότι οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την επίτευξη στόχων που θα επιτρέψουν να υπάρξει βελτίωση μεγαλύτερη από το αν χρησιμοποιηθούν μονάχα, αν μάλλον δαπανηθούν μονάχα τα χρήματα στο επίπεδο των χωρών μελών. Διότι χώρες μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί μπορούν ίσως να συγκεντρώσουν επαρκή κονδύλια στον τομέα αυτό αλλά δυστυχώς λόγω των του κατακαιρματισμού των προσπαθειών δεν είμαστε σε θέση να ανταγωνιστούμε άλλες χώρες όπως οι Ενωμένε Πολιτείε, όπως η ε, Κίνα ή οι Ινδίες. Ενώ εάν συμπαραταχθούμε, εάν εμφανιστούμε ενωμένοι μπορούμε να επιτύχουμε πολύ περισσότερα. Το μέγα ερώτημα που τίθεται όμως είναι το εξής. Είναι πράγματι διατεθειμένες οι χώρες μέλη να παρετηθούν από την ιδέα ότι θα χρηματοδοτούν οι ίδιες και θα ρυθμίζουν οι ίδιες τις πολιτικές τους εκπαίδευσης, έρευνας. Αντιλαμβάνονται ότι εδώ ισχύει το, η ισχύ τη ενώση. Η δεύτερη μου παρατήρηση αναφέρεται στο κλείσιμο των πυρηνικών σταθμών. Θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι Εάν διαθέσουμε κονδύλια για το κλείσιμο των πυρηνικών εργοστασίων, θα πρόκειται για πυρηνικά εργοστάσια τα οποία αποτελούν κάποιο κίνδυνο ε, υπό την παρούσα κατάσταση λειτουργίας τους και όχι μόνο για την χώρα μέλος στην οποία είναι εγκατεστημένα αλλά και για τις υπόλοιπες. Αυτό θα δικαιολογούσε μια τέτοια κίνηση και θα πρέπει για αυτό να ε, διατεθούν κονδύλια και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον προϋπολογισμό μας έχουμε κονδύλια τα οποία προβλέπονται να δαπανηθούν και για την πρόθεση ανανεώσιμων ενεργειών. Εγώ όμως θα ήθελα να διαχωριστούν αυτοί οι δύο τομείς. Διότι εδώ υπάρχει, υπάρχουν και σοβαρές αποκλίσεις απόψεων σε ό,τι αφορά την πυρηνική ενέργεια. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που θεωρούν ότι η πυρηνική ενέργεια είναι άκρος επικίνδυνη και ότι η εγκατάληψή της είναι μονόδρομος. Υπάρχουν όμως και άλλοι που θεωρούν ότι δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα παρά μόνο να διατηρήσουμε αυτήν την τεχνολογία. Στον τομέα ωστόσο των ανανεώσιμων ενεργειών και γι' αυτό είμαι βέβαιος θα χρειαστεί να διαθέσουμε περισσότερα κονδύλια και από τις χώρες μέλη για την επίτευξη πρόοδου. Σας ευχαριστώ αγαπητέ φίλε. Ξανάρχομαι στα Εθνικά Κοινοβούλια. Η κυρία Αλίσια Κολιτσόφσκα της Πολωνικής Βουλής. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, η Πολωνία εξακολουθεί να πιστεύει ότι είναι πολύ σημαντικό και για την Πολωνία και για τον κοινοτικό προϋπολογισμό η συνέχιση της πολιτικής συνοχής. Η πολιτική συνοχής συνδυάζεται φυσικά με την ανάπτυξη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Κάθε χώρα μέλος θα έπρεπε να προβεί σε μια ιεράρχηση των επιλογών και των προτεραιοτήτων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των περιφερειών της των περιφερειών του κάθε κράτους και με βάση φυσικά και τη στρατηγική του 2020. Σίγουρα θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στα συνθήματα της καινοτομίας, της ανάπτυξης των υποδομών, στις ε, υποδομές των μεταφορών, των επικοινωνιών, αλλά και στην ανάπτυξη της ευρηματικότητας, της δημιουργικότητας και του πολιτισμού. Οι περιφέρειες χρήζουν ιδιαίτερης υποστήριξης και μάλιστα ιδιαίτερα οι περιοχές που υπέστησαν σημαντική υποχώρηση στην ανάπτυξή τους εξαιτίας οικονομικής κρίσης. Σημαντικό ρόλο στην πολιτική συνοχή θα πρέπει να εξακολουθεί να διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι συζητήσεις για τον τρόπο χρηματοδότησης του κοινοτικού προϋπολογισμού. Το σημερινό σύστημα των ιδίων πόρων πολύ συχνά θεωρείται κάπως αδιαφανές και ιδιαίτερα περίπλοκο η συζήτηση για τον κοινοτικό προϋπολογισμό θα πρέπει να καλύψει και τις δομές του προϋπολογισμού και όχι όπως συνήθως να περιορίζεται στον όγκο του προϋπολογισμού, στο μέγεθος και τις διαστάσεις του. Τα ενδεχόμενοι νέοι ειδηπόροι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να λαμβάνουν υπόψη την αρχή της ισοτιμίας των υποχρεώσεων και της δικαιοσύνης και φυσικά να έχουν σχέση με την δυνατότητα της κάθε χώρας για τη συμβολή στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Καλό θα ήταν να επικεντρωθούμε σε γενικές συζητήσεις. Γίνονται προτάσεις για ένα κοινοτικό φόρο, γίνονται προτάσεις για νέες πηγές ε, του κοινοτικού προϋπολογισμού, για παράδειγμα έσοδα από την πώληση των δικαιωμάτων εμπορίας ε, των εκπομπών, είναι συζητήσεις και προτάσεις που θα μπορούσαν να διαρευνηθούν. Είναι πιθανές ε, νέες πηγές του κοινοτικού προϋπολογισμού και εξετάζονται και από το δικό μας Υπουργείο Οικονομικών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Βούτερς της Βελγικής Βουλής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μια και το θέμα του συντονισμού και της ε, συνέργειας μεταξύ του κοινοτικού προπολογισμού και των εθνικών προπολογισμών ε, βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης, θα ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι και εγώ τις ανησυχίες και τους ενδιασμούς ως προς την ε, ελλειπή διαβούλευση που προβλέπεται στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Εμείς αντιμετωπίζουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή με την έλλειψη κυβέρνησης, αλλά δεν αποκλείεται και άλλες χώρες να βρεθούν σε αντίστοιχη κατάσταση, γιατί όταν διεξάγονται εκλογέ σε μια χώρα, αυτό που με ανησυχεί είναι ότι η κυβέρνηση προσδιορίζει την δημοσιονομική πολιτική για την επόμενη τετραετία. Και φυσικά υπάρχουν διάφορες επιλογές πολιτικής που γίνονται, κάτι που διαμορφώνει και καθορίζει και την οικονομική και κοινωνική πολιτική μιας χώρας. Ερωτώ λοιπόν το εξή. Τι συμβαίνει στις άλλες χώρες. Γνωρίζω ότι δεν υπάρχει υποχρέωση και μπορεί σε άλλες χώρες τα εθνικά κοινοβούλια να εμπλέκονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης που θα υποβληθεί στα τέλη Μαρτίου και άκουσα την κυρία Μπέρες που λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει λόγο, αλλά θα ήθελα να ακούσω και τις απόψεις των άλλων χωρών. Πώς έγιναν οι διαβουλεύσεις στα υπόλοιπα Εθνικά Κοινοβούλια, γιατί είναι σημαντικό τα κοινοβούλια να δίνουν τη γνώμη τους, να συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις. Γιατί έτσι καθορίζεται η οικονομική και κοινωνική πολιτική μιας χώρας. Πώς είναι δυνατόν να γίνεται ερήμην του Εθνικού Κοινοβουλίου μια τέτοια πολιτική γιατί στη συνέχεια οι βουλευτές καλούνται να τηρήσουν κάποιες υποσχέσεις που είχαν δοθεί και κάποιες δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν. Είπατε ότι τον Ιούνιο οι Υπουργοί Κοφίν και οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων θα εξετάσουν και θα κρίνουν τους υπόλοιπους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αυτό για μένα είναι αρκετά αφιλεγόμενο. Ποιο είναι ο βαθμός αντικειμενικότητας σε ό,τι αφορά την ανάλυση αυτών των προπολογισμών. Γιατί μπορεί κανεί να πει για, ένα για έναν εθνικό προπολογισμό ότι δεν είναι ικανοποιητικό. Αλλά αυτό είναι σαν να μπαίνει στο δόλιο του κατηγορουμένου μια χώρα. Και πώς αντιδράσουν οι χρηματοπιστωτικέ αγορέ απέναντι σε μια τέτοια κρίση. Πώς είναι δυνατόν 27 Υπουργοί Εκοφήν να προβούν σε αξιολογικές κρίσεις που ίσως έχουν ολέθριες συνέπειες για συγκεκριμένες χώρες. Τι θα γίνει αν 27 υπουργοί θεωρήσουν ότι οι προσπάθειες που κάνει μια χώρα για να εξηγιάνει τα οικονομικά της είναι ανεπαρκή. Μια τέτοια κρίση θα έχει σοβαρές συνέπειες για την φήμη αυτής της χώρας και αντίκτυπο στην εικόνα της στις χρηματαγορές. Στο Βέλγιο υπάρχουν κάποιες πολιτικές που δεν αποτελούν πλέον εθνική αρμοδιότητα, αλλά περιφερειακή. Οι αποφάσεις λαμβάνονται σε περιφερειακό επίπεδο και οι περιφερειακές βουλές είναι ακόμη πιο απούσες από τον μηχανισμό αυτό. Όταν μιλούμε για καινοτομία, έρευνα, ενέργεια, μιλούμε για αρμοδιότητες που σε πολλές χώρες μέλη εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των περιφερειακών βουλών. Πώς εξασφαλίσουμε η συμμετοχή και των περιφερειακών κοινοβουλίων στην όλη αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. πρόεδρες Μότα Πίντου από την Πορτογαλική Βουλή. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να υπενθυμίσω ότι αυτή είναι η πρώτη χρονιά της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που δεν ήταν μια καθόλου εύκολη χρονιά για τη χώρα μου. Είναι γνωστό αυτό. Και παρόλο που αυτό φυσικά δεν έχει σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, η κατάσταση στην Πορτογαλία, είναι αλήθεια το πρόβλημα συντονισμού των εθνικών προπολογισμών και μια κάποια δυσκολία ή έλλειψη συντονισμού στην υποβολή των προτάσεων που συζητήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ακριβώς επειδή δεν εξετάστηκαν αυτές οι προτάσεις στην Πορτογαλία πριν παρουσιαστούν στο Συμβούλιο, αυτό οδήγησε στην πολιτική κρίση που το Μάρτιο ανέτρεψε την κυβέρνηση της Πορτογαλίας. Βέβαια, η σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι πολύ αδύναμη, αλλά απλώς ήθελα να το επισημάνω. Θα ήθελα επίσης να πω ότι αυτή τη χρονιά η κρίση έφτασε και στην Πορτογαλία. Η Πορτογαλία επλήγει από το συσσωρευμένο αποτέλεσμα των ανισορροπιών και τη διόγκωση του δημόσιου χρέους, δημόσιου χρέους της. Αλλά η κατάσταση αυτή που δεν πλήττει μόνο την Πορτογαλία αλλά και άλλες ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα γενικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει μια εύκολη εξήγηση ή μια θαυματουργή λύση για την εξυγίαση των δημόσιων οικονομικών. Ούτε μπορούμε να κατηγορήσουμε μόνο το χρηματοπιστωτικό τομέα, μόνο τις τράπεζες. Το πρόβλημα έγκυται στην έλλειψη αξιοπιστίας των εθνικών λογαριασμών στις περισσότερες χώρες και οι πορτογαλικές οικονομικές δυσκολίες ε, μας επαναφέρουν στο, στο πρόβλημα των ε, νομισματικών ζωνών, ίσως ε, και μας δημιουργεί προβληματισμό για το κατά πόσο έγιναν σωστές προσπάθειες για την εφαρμογή του ευρώ ή δόθηκε αρκετή σημασία στην ανάπτυξη στα πλαίσια της προσπάθειας της προσαρμογής και στο ευρώ. Η λύση τελικά που υιοθετήθηκε ελπίζω να γίνει δεκτή και ελπίζω να συγκεντρωθεί η πολιτική υποστήριξη για το πρόγραμμα της δημοσιονομικής εξυγίασης και στην Πορτογαλία. Πρώτη, πρώτα θέλουμε την εξυγίαση των δημοσίων οικονομικών και μετά την ελάφρυνση του χρέους και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα μας επαναφέρουν και πάλι στον δρόμο της ανάπτυξη. Βέβαια, η σημερινή συζήτηση εδώ επικεντρώνεται κυρίως στο θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Και όπως σας είπα, ο βασικός λόγο για τον οποίο απορρίφθηκαν στην Πορτογαλική Βουλή τα μέτρα που υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι γιατί δεν είχαν συζητηθεί προηγουμένω πριν την παρουσίαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν είχαν συζητηθεί αρκετά στην Πορτογαλία και αυτό οδήγησε στην απόρριψή του. Η διαπραγμάτευση όλων αυτών των μέτρων ναι, έγινε λίγο παρασκηνιακά και κλεισμένο των θυρών, χωρί προηγούμενη συζήτηση. Κάτι που οδήγησε στην απόρριψή του. Βέβαια, ίσω η διαδικασία αυτή ε, οφειλόταν στον επίγοντα χαρακτήρα τη κατάσταση, αλλά θέλουμε να, απο, να αποτραπεί μια επανάληψη τέτοιας α, κρυψίνιας στο μέλλον. Μιλήσατε κύριε Λαμασούρ και για το σχέδιο σταθερότητας και ανάπτυξης και το θέμα της επικαιροποίηση των αιτήσεων σχεδίων σύγκλησης και σταθερότητας και τα κατά πόσο θα πρέπει να υποβάλλονται αυτά τα σχέδια πριν ή μετά τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υποβάλλονται αυτά τα σχέδια σύγκλησης και σταθερότητα μετά του εθνικού προπολογισμού ώστε οι προβλέψεις για το επόμενο έτος να στηρίζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό. Μια άλλη εναλλακτική λύση που προτάθηκε ήταν η πρόταση αν τα μέτρα ή προτινόμενοι στόχοι κρυθούν ανεπαρκή, το κράτος μέλος να μπορεί να τους τροποποιήσει αυτούς τους στόχους και τα μέτρα το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, όταν θα εγκρίνει τον εθνικό του προϋπολογισμό. Ανακύπτει όμως το ερώτημα, σε ποιο βαθμό έτσι περιορίζονται de facto οι αρμοδιότητες των Εθνικών Κοινοβούλων εφόσον δεν διδραματίσουν κανένα ρόλο στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Γιατί τελικά αποσυνδέεται η Εθνική Βουλή, κάθε, το κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και δεν συμμετέχει στο πράσινο φως που δίνεται σε αυτή τη διαδικασία και στον ετήσιο προπολογισμό συγκεκριμενοποιούμε τον πολιετή προγραμματισμό και τους προσανατολισμούς των προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκληση, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ανάμειξη των εθνικών κοινοβουλίων στο καθορισμό και το μεσοπρόθεσμο στρατηγικών. Θα πρέπει να υπάρχει μια, καλύτερη προετοιμασία των γενικών γραμμών του προϋπολογισμού και επίσης καλύτερη συμμετοχή και ανάμεξη σε προγενέστερο στάδιο των Εθνικών Κοινοβουλίων για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Για να μην ε, εμφανίζονται μόνο σε μεταγενέστερο στάδιο της ε, διαδικασίας και επαναληφθεί αυτή η δυσαρέσκεια των Εθνικών Κοινοβουλίων που δεν ε, έδωσαν το λόγο τους, που δεν εισακούστηκε η φωνή τους, γιατί οι διαπραγματεύσει έγιναν ερήμην τους από τις κυβερνήσεις της Βρυξέλλες. Ευχαριστούμε Πρόεδρε. Πήραμε το μήνυμα σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ σε μια στιγμή όπου η χώρα σας αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες και όπου σύντομα θα έχετε και βουλευτικές εκλογές. Επανερχόμεθα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την κυρία Τρούπελ. Ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο. Θα παρέμβω σύντομα θυμίζοντας κάτι που είχε πει ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ «I have a dream» Έχω ένα όραμα και χαίρομαι που διεξάγουμε την κοινή αυτή συνάντηση εδώ βουλευτών από πολλές χώρες μέλη και ε, μεταξύ αυτών δηλαδή και ημών που είμαστε από διάφορους πολιτικού σχηματισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διότι θεωρώ ότι μας δίνει μια καλή ευκαιρία και ότι είναι πραγματικά χρόνος να καθορίσουμε ποια είναι τα κοινά μας ε, συμφέροντα. Διότι έχουμε συνηθίσει να βρισκόμαστε σε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι το ευρωπαϊκό επίπεδο κατά των εθνικών επιπέδων, οι κακές Βρυξέλλες. Αυτό όμως είναι πρόβλημα εάν συνεχίσουμε να παίζουμε το παιχνίδι αυτό, διότι από την πολιτική σκοπιά θα σημαίνει ότι αποτυγχάνουμε στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι πάντοτε χρήσιμο να προσπαθούμε να εντοπίσουμε κοινά συμφέροντα, να εξετάζουμε την παγκόσμια κατάσταση και αν εμείς στην Ευρώπη δεν κατανοήσουμε ότι οφείλουμε να συνεργαστούμε για να είμαστε ισχυροί στον παγκόσμιο ανταγωνισμό με τις Ηνωμένε Πολιτείε, την Ινδία, την Κίνα, την Βραζιλία. Βρίσκω ότι τότε θα αντιμετωπίσουμε μεγάλο κίνδυνο τελικά να αποτύχουμε, να είμαστε εμεί οι χαμένοι. Μπορούμε να εντοπίσουμε κοινά συμφέροντα. Πρόκειται κυρίως για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ως μέλος της ομάδας των πράσινων, ανταγωνιστικότητα σημαίνει σήμερα ότι οφείλουμε να την συνδυάσουμε και με προηγμένη τεχνολογία οικολογικού χαρακτήρα που θα προσφέρει και απασχόληση νέα προϊόντα για την εσωτερική ενιαία αγορά αλλά και για την παγκόσμια αγορά. Και όταν μιλούμε για τη στρατηγική της Ευρώπης του 2020 στο εθνικό επίπεδο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε κοινά συμφέροντα να επενδύσουμε περισσότερο στην παιδεία, την εκπαίδευση, την έρευνα, την ανάπτυξη, οι δεν θα είμαστε έτοιμες και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον νέο ανταγωνισμό. Και εάν παραβλέψουμε τα συμφέροντά μας στην πολιτική συνοχή και στην γεωργία, εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις όπως αλλαγή του κλίματος, ε, βιωσιμότητα και της ανάπτυξης, πρέπει να αναδιαμορφώσουμε και την αγροτική πολιτική και την πολιτική συνοχής με τρόπο πιο αηφόρο. Άρα θα έχουμε μεγάλα τμήματα του κοινοτικού προϋπολογισμού και τμήματα των εθνικών προϋπολογισμών που θα πρέπει να εξυπηρετούν κοινού στόχους. Θα έλθω τώρα στο θέμα των ιδίων πόρων του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Γνωρίζω ότι είναι θέμα ευαίσθητο και δύσκολο να πιστούν οι διάφορες πλευρές. Αλλά επιτρέψτε μου να θέσω υπόψη σας τα επιχειρήματά μου, για ποιο λόγο δηλαδή θεωρώ ότι ευρωπαϊκοί ήδη πόροι, όπως για παράδειγμα φόρος επί της κυροζήνης ή φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, θα μπορούσαν να σημάνουν μια πολύ καλή συμβολή στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, γιατί όλα αυτά τα αντικείμενα φορολόγησης έχουν διαμεθοριακό χαρακτήρα και θα κατανοήσουν οι πολίτες εν τέλει ότι μπορεί να είναι μια καλή ιδέα διότι από την αρχή, από την απαρχή των ευρωπαϊκών συνθήκων οι ίδιοι πόροι είναι κατοχυρωμένοι στις συνθήκες. Δεν πρόκειται για νέα ιδέα. Πρέπει όμως να τις εμφυσίσουμε νέα ζωή. Γι' αυτό νομίζω ότι ό,τι και αν συζητήσουμε στο τεχνικό επίπεδο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού Κυρίως πρόκειται ωστόσο για το πολιτικό θέμα, αν υπάρχει δηλαδή εμπιστοσύνη μεταξύ μας και η πολιτική βούληση να κάνουμε προσπάθεια εξασφάλισης και ε, να δώσουμε μια νέα όθηση στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Γιατί αν δεν κάνουμε κοινή προσπάθεια το ευρωπαϊκό και τα εθνικά επίπεδα θα αποτύχουμε. Γι' αυτό με την ευκαιρία της σημερινής συνάντησης ζητώ τουλάχιστον να συμφωνήσουμε στο τι διακυβεύεται. Και όπως είπα στην αρχή της ομιλίας μου, ξαναλέω, έχω ένα όραμα. Ευχαριστώ, Έλγα, λέει ο, ο ε, πρόεδρος Λαμασούρ. Βρίσκεται κοντά μας εκπρόσωπος της Λιθουανικής Βουλής, ο κύριος Ανδρουκάητης. Gerbiamas για το Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς στη Λιθουανία έχουμε ισχυρή βουλή και η βουλή αυτή έχει Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων όπου Στις συναντήσεις με αυτήν συμμετέχουν και πρόεδροι άλλων επιτροπών, όπως ε, της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Βουλής μας. όπου σχεδιάζουμε διάφορα προγράμματα, καθώς και κάνουμε τον ετήσιο προγραμματισμό μας, καθώς και το συντονισμό με το πρόγραμμα σύγκλησης. Φέτος Έχουμε εκτελέσει τα καθήκοντά μας εν ώψη και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, έχουμε κάνει τη σχετική προετοιμασία, έχουμε διεξαγάγει συζητήσεις για τις κατευθυντήριες γραμμές των εθνικών προγραμμάτων, για τις παραμέτρους που πρέπει να επιδιώξουμε να εφαρμόσουμε μέχρι τέλους του έτους. Τώρα αναμένουμε την λήψη μέτρων από την κυβέρνηση. Μετά από την συζήτηση στην Επιτροπή μας αναμένουμε λοιπόν το σχέδιο προγράμματος της κυβέρνησης. Βέβαια, συμμετέχουμε στην Ευρώπα ΣΥΝ, δεν είμαστε μέλος της Ευρωζώνης, αλλά λαμβάνουμε μέτρα συντονισμού της φορολογικής μας πολιτικής και ασφαλώς κάνουμε προσπάθεια να προσεγγίσουμε την Ευρωζώνη με σταδιακή προσαρμογή μας στα κριτήρια της Κοπενχάγης. Το 2008 είχαμε προσεγγίσει ήδη πάρα πολύ. Πρόκειται για λίγες θέσεις μετά την υποδιαστολή στην πραγματικότητα ε, για τις οποίες αποτύχαμε και βεβαίως η οικονομική κρίση που επήλθε μετά μας απομάκρυνε περισσότερο από τον στόχο αυτό. Βέβαια, Ασφαλώς έχουμε ένα αυστηρό πρόγραμμα εξοικονομήσεων στον δημόσιο τομέα. Έχουμε περικόψει σημαντικότατα τις δαπάνες, κάτι το οποίο προκάλεσε κοινωνικές εντάσεις στη χώρα μας. Αλλά λάβαμε και άλλα μέτρα. Επιδιώκουμε τους στόχους μας και σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τον συντονισμό των ε, δημοσιονομικών και οικονομικών πολιτικών, όλες οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούνται μεταξύ αυτών και την εισαγωγή πρόσθετων φορολογιών και τα θέματα επίσης των πρόσθετων ίδιων πόρων. Ωστόσο είναι πολύ εκτεταμένη αυτή η συζήτηση. Δεν αρκούν μόνο οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στον τομέα του συντονισμού των δημοσιομικών πολιτικών οφείλουμε ακόμη να συζητήσουμε πολύ και ε, η ατζέντα είναι ευρύτατη. Τελευταίος κ. Βούντερ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει το λόγο μετά από τον κύριο Μίλντερ θα κλείσουμε με τα συμπεράσματα. Δεν θα κάνω εγώ αυτή τη δουλειά, αλλά εν πάση περιπτώσει σχετικά με αυτά τα οποία είπε και η Χέλγα Τρούπελ. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που είναι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου με τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νομίζω ότι μαζί εμείς μπορούμε να αποφασίζουμε, να παίρνουμε αποφάσεις για τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε τίποτα να πούμε για τους ιδίους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δείτε τα τελευταία χρόνια αυτό είναι το βασικό θέμα που συζητιέται. Δεν νομίζω πως σε αυτή τη φάση μπορούμε να θεωρούμε πάντα πως για μία χώρα από το 1984 ισχύει ένας ειδικό κανονισμός, ο οποίος λέει ότι ό,τι πληρώνει η χώρα αυτή πρέπει να παίρνει πίσω κατά τα δύο τρίτα τη διαφορά. Αν ισχύει κάτι τέτοιο θα πρέπει να το εφαρμόσουμε για όλες τις χώρες που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Η συνθήκη της Λισαβόνας άλλωστε διευκρινίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει ιδίους πόρους. Από την αρχή της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας αυτό έχει ερμηνευθεί όχι όπως ερμηνεύεται τώρα με άμεσες συνεισφορές των κρατών μελών, αλλά μια ανεξάρτητη εισοδηματική πηγή. Αυτό θα το αποφασίσουν τα, εθνικά κοινοβούλια. Το σύστημα το οποίο έχουμε τώρα είναι πλήρως ακατανόητο, είναι στρεβλό, και σαν μέλος δεν το καταλαβαίνω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και νομίζω ότι δεν υπάρχουν καν υπάλληλοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι οποίοι να ελέγχουν απόλυτα το θέμα. Είναι πολύ περίπλοκο το σύστημα, πρέπει εμείς να ξεφύγουμε από την αντίληψη αυτή. Από το 52 μέχρι το 90 είχαμε άλλωστε ένα σύστημα το οποίο βασιζόταν σε ανεξάρτητους ε, ιδίους πόρους εν μέρη από υπάρχοντες φόρους. Δεν βρίσκω το λόγο γιατί να μην αναζωογονήσουμε το συγκεκριμένο αυτό παλαιό σύστημα και να ξεφορτωθούμε όλα τα αρνητικά σχόλια για τους ευρωπαϊκούς φόρους. Κανένας δεν θέλει να επιβάλλει νέους ευρωπαϊκούς φόρους. Αυτό που θέλουμε είναι να υπάρξει ανεξάρτητο εισόδημα από τους υπάρχοντες φόρους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ συνάδελφε Μιλντά. Καλώς. Νομίζω ότι έχει έρθει η στιγμή για να κλείσουμε τις εργασίες μας. Δεν θα ήθελα να βγάλω συμπεράσματα, αλλά να σας προτείνω μια διαδικασία για να ακολουθήσουμε από εδώ και πέρα. Όλοι συνειδητοποιούμε ότι βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση. Είμαστε κατεστραμμένοι. Αυτό έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Μας υποχρεώνει να φανούμε εφάνταστοι και θαραλέοι. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση λοιπόν όπου ορισμένες χώρες πηγαίνουν πιο άσχημα από άλλες και έχουν ανάγκη από τη βοήθεια των υπολείπων. Στην δυστυχία λοιπόν, την συνολική δυστυχία, η ευρωπαϊκή οικογένεια υπάρχει και έχουμε θέσει αυτούς στόχους και για να μπορέσουμε να βγούμε από την ασθένεια η οποία μας κυνηγά αλλά και να προετοιμάσουμε το μέλλον. Πώς θα μπορέσουμε με τον καλύτερο τρόπο να συνεργαστούμε, αυτό έχει σημασία. Αυτό ήταν και ο στόχος αυτής της συνάντησης και σας ευχαριστώ για τις ιδέες σας πολύ συγκεκριμένες και πολύ θετικές. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα από εδώ και πέρα. Την 20 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει την πρότασή της την επόμενη εβδομάδα με το σχέδιο προϋπολογισμού της Ένωσης για το 12. Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο προϋπολογισμός. Κάνω μία πρόβλεψη παρακινδυνευμένη ότι θα υπάρξει μια ελάχιστη αύξηση ή ίσως και μια μείωση ελάχιστη. Αυτό σας κάνει να γελάτε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα δούμε πώς θα γελάσετε την επόμενη εβδομάδα. Στη συνέχεια σε διάφορα κοινοβούλια θα γίνουν κάποιες συζητήσεις δημοσιονομικές. Ο καθένας προετοιμάζει το εθνικό του πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης. Την 29η Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει μία πρόταση την ίδια στιγμή για πρώτη φορά και τις προτάσεις της για το δημοσιονομικό πλαίσιο το πολιετές, το επταετές συγκεκριμένα, για τον κοινοτικό προϋπολογισμό, γι' αυτό μιλάμε, 2014-2020. Και θα κάνει και μία πρόταση για τους πόρους, για τα έσοδα. Πολλοί συναδέλφοι αναφέρθηκαν στα έσοδα που χρηματοδοτούν τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ποιος χρηματοδοτεί σήμερα, εσείς οι φόροι που εσείς αποφασίζετε να δώσετε στην Ένωση. Και αυτό γίνεται κάτω από συνθήκες αρκετά θα έλεγα σκοτεινές. Δεν είναι αυτό το θέμα μας όμως σήμερα. Είναι όμως παρόλα αυτά ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει πέρυσι και θα πρέπει να επανέλθουμε και τον επόμενο χρόνο. Την 29η Ιουνίου λοιπόν όλα αυτά θα δημοσιοποιηθούν να ποιες είναι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών για το πρόγραμμα της Ευρώπης 2020 αλλά και για τις άλλες πολιτικές της Ένωσης, της αναπτυξιακής βοήθειας, της εξωτερικής πολιτικής, της ΚΑΠ κτλ. Το φθινόπωρο σε όλα τα κοινοβούλια θα ψηφιστεί ο ετήσιος προϋπολογισμός και ταυτόχρονα οι Υπουργοί Οικονομικών όταν συνεδριάσουν στα πλαίσια αυτού που ονομάζουμε κοφίν, αλλά και το Συμβούλιο θα ολοκληρώσουν την διαμόρφωση των διαδικασιών για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει συνεισφέρει σε αυτή τη συζήτηση με την έκθεση της κυρίας Μπερές, η οποία ήταν παρούσα εδώ και η οποία άκουσε προσεκτικά αυτά που είπατε και η οποία θα τα λάβει υπόψη. Και υποθέτω, υποθέτω ότι σε κάθε μία από τις χώρες μας θα υπάρξει μία διαπραγμάτευση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο για να δούμε πώς κάθε κυβέρνηση θα συνεργαστεί με την Βουλή της για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Διάβασα σε ορισμένες εφημερίδες ότι έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις σε ορισμένες χώρες. Κάποιοι αναφερθήκατε σε αυτές τις, ε, τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο νομοθετικό και το εκτελεστικό στη χώρα σας. Αυτά θα γίνουν κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου, λοιπόν, του ενεστώτος έτους. Μου φαίνεται ότι αυτό το οποίο θα ήταν χρήσιμο κατά τη διάρκεια αυτού του δευτέρου εξαμήνου, μιλάμε για το 11, είναι να υπάρξει ένα παρατηρητήριο θα έλεγα του τι συμβαίνει σε κάθε χώρα και σε κάθε εθνικό κοινοβούλιο γύρω από την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Το πρώτο θα έλεγα ουσιαστικό Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα είναι το πρώτο του 2012. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του δεύτερου μισού του 2011 θα είμαστε κάτω από Πολωνική Προεδρία και αυτό προτείνω είναι σε συνεργασία με τους Πολωνούς φίλους να δούμε πώς μπορούν να οργανώσουν ή από κοινού να οργανώσουμε αυτό το παρατηρητήριο θα έλεγα, έτσι ώστε να συλλέξουμε τις πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από όλες τις χώρες και από όλα τα κοινοβούλια, για να δούμε πόσο καθένας θα μπορέσει να οργανώσει τη συμμετοχή του στην προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Στη συνέχεια θα φτάσουμε στις αρχές ε, του 12, σε ένα σχεδόν χρόνο. Εκεί το θέμα το οποίο πρέπει να θέσουμε νομίζω, νομίζω, θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα στις αρχές του επόμενου χρόνου να υπάρξει μια πραγματική συνάντηση εκπροσώπων των Επιτροπών Οικονομικών των Κοινοβουλίων των Κρατών Μελών για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε τη συζήτηση. Μην περιοριζόμεθα όπως σήμερα μόνο σε κάποιες γενικού τύπου παρατηρήσεις, διαδικαστικού περισσότερο τύπου, αλλά παρατηρήσεις οι οποίες άπτονται της ουσίας, και μάλιστα επί τη βάση των εγγράφων τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέσει υποδιαβούλευση στις αρχές του πρώτου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ε, θέματα όπως οι προοπτικές ανάπτυξης και τα βασικά χαρακτηριστικά της εξέλιξης της ευρωπαϊκής οικονομίας που θα πρέπει να δημοσιεύσει τον μήνα Ιανουάριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 12. Ανάμεσα στον Ιανουάριο του 12, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει τις οικονομικές της υποθέσεις, τα σενάρια της, και στο τέλος Μαρτίου, όπου θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο καθορίζει τους βασικούς προσανατολισμούς, είναι προφανές ότι σε κάθε μία από τις χώρες μας θα γίνει μια εθνική συζήτηση. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να γίνει μια τέτοια συνάντηση κάτω από την δανική αυτή τη φορά προεδρία. Το λέω αυτά μπροστά στους εκπροσώπους του Folketing είτε με την Προεδρία του Φόλκετιν, είτε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, δεν έχει αυτό σημασία. Αλλά θα μπορούσαμε να συναντηθούμε λοιπόν στις αρχές του εξαμήνου αυτού για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα αντιδράσουμε σε αυτά τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλωστε, στις ανταλλαγές απόψεων και στις συζητήσεις μας, θα πρέπει να τεθεί επίσης και το θέμα του περιεχομένου του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, Πολλοί από εσά είπατε ότι ο καθένας θα πρέπει να κάνει προσπάθειες και εμείς κάνουμε προσπάθειες. Θα πρέπει και το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο να κάνει προσπάθειες οικονομία, εξοικονόμηση, στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Είναι λογικό αυτό. Εσείς τον χρηματοδοτείτε. Οι Υπουργοί Οικονομικών σας. Ταυτόχρονα, εμείς θα προσπαθήσουμε όταν προχωράμε στις δαπάνες, οι δαπάνες αυτές ε, να χρηματοδοτούν τις μελλοντικέ πολιτικές. Πολλοί από σας είπατε ότι θεωρούμε ότι ο προπολογισμό πηγαίνει πάρα πολύ στη Γεωργία. Άλλοι είπατε ότι θέλουμε να κάνουμε περισσότερα για κάποιες υποδομές και να υπάρχουν λιγότερες δαπάνες. Οι Υπουργοί Προϋπολογισμών σας τα διευκρινίζουν αυτά. Αλλά καλό θα είναι να τα συζητήσουμε και μεταξύ μας, έτσι ώστε μετά από αυτή την ανταλλαγή απόψεων, ο καθένας να μπορέσει στα πλαίσια της εθνικής συζήτησης της δημοσιονομικής να θέσει και τα ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά του θέματος. Δεν είμαστε μόνοι μας, υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι μπορούν να με βοηθήσουν είτε άμεσα είτε έμεσα και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη μας καλύτερα τις εθνικές ανησυχίες έχοντας μια αντίληψη η οποία να μην είναι η αντίληψη της δίκαιης επιστροφής, δηλαδή όσα δίνεις τόσα παίρνεις, αλλά μια συνεκτική αντίληψη που λέει αυτά τα λίγα χρήματα πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα για τη χώρα μου και γενικότερα για την ευρωπαϊκή οικογένεια. Εφόσον μπορούμε να οργανώσουμε μια τέτοιου τύπου συνάντηση και εφόσον πετύχει μια τέτοια συνάντηση και θεωρήσουμε ότι είναι ενδιαφέρουσα και μπορεί να είναι ένα χαρακτηριστικό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, είναι κάτι το οποίο μπορεί να επαναληφθεί. Αυτό το οποίο καταλάβαμε όλοι νομίζω είναι ότι στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να προσπαθήσει να είναι χρήσιμο προς όλους. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι αυτού του τύπου οι συναντήσεις είναι χρήσιμες, έστω και σε αιτήσια βάση, τότε σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε να αρπάξουμε την ευκαιρία για να μπορέσουμε να συζητήσουμε μεταξύ μας το πολιετές πλαίσιο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και το θέμα της πολιετούς του χρηματοδότησης. Ένα θέμα επί του οποίου αυτή τη στιγμή υπάρξει μια τέτοια συμφωνία, εσείς είστε που θα το αποφασίσετε, εσείς στα κοινοβούλια των κρατών μελών έχετε την τελευταία λέξη. Όσο όμως περισσότερο συνεργαστούμε και όσο νωρίτερα συνεργαστούμε, τόσο θα επηρεάσουμε θετικά το τελικό αποτέλεσμα. Πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο θέμα της χρηματοδότησης του κοινοτικού προϋπολογισμού. Σήμερα χρηματοδοτείται από τις εθνικές συνεισφορές. Ο συνάδελφος Γιάν Μούλντερ είπε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει λόγο στο τμήμα των εσόδων αλλά να προσθέσω εδώ ούτε κι εσείς έχετε λόγο. Κανένας δεν έχει να συζητήσει το θέμα των εθνικών συνεισφορών. Για τα κράτη-μέλη πρόκειται για μια υποχρεωτική δαπάνη. Τα κοινοβούλια λοιπόν των κρατών μελών ψηφίζει, ψηφίζουν τις εθνικές τους συνεισφορές, αλλά στην ουσία είναι μία ψήφος υποχρεωτική. Δεν μπορείτε να μειώσετε ούτε κατά τα ένα ευρώ τη συνεισφορά την εθνική. Αυτά προβλέπουν οι συνθήκες, αυτά αποφασίζονται και κλεισμένων των θυρών από τους υπουργού οικονομικών και από τους υπαλλήλους που κάνουν μαθηματικούς υπολογισμούς και πράξεις και χρειάστηκαν εννέα σελίδες στην τελευταία επίσημη εφημερίδα για να περιγραφεί η εθνική συνεισφορά. Λοιπόν είναι παράλογη η μέθοδος αυτή, είναι αντιδημοκρατική η μέθοδος αυτή. Δεν υπάρχει έστω και ένας βουλευτής, εθνικός ή ευρωβουλευτής που να είναι σε θέση να πει γιατί η εθνική συνεισφορά της χώρας από την οποία προέρχεται είναι καθορισμένη στο επίπεδο στο οποίο είναι καθορισμένη. Κανείς δεν μπορεί να το δικαιολογήσει αυτό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και αυτό είναι ένα θέμα επί το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Οι ευρωπαϊκοί προϋπολογισμοί κοστίζουν. Εσείς πληρώνετε και εμείς εποφελούμεθα. Επ' αυτού μέχρι τώρα δημόσια συζήτηση δεν έχει γίνει. Το συζητάμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά στα κράτη-μέλη συζήτηση δεν γίνεται. Αυτό περιορίζεται σαν συζήτηση σε ένα κλειστό αριθμό, σε ένα κλειστό κύκλο υπουργών οικονομικών και συνεργατών. Αυτό πρέπει να τελειώνει πια. Μετά από τις κρίσεις οι οποίες προκλήθηκαν και στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σε κάθε χώρα, όπου είμαστε υποχρεωμένοι να δαπανάμε λιγότερα και καλύτερα, είναι σαφές ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια νέα μέθοδο χρηματοδότησης. Όλοι είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες, όλοι είμαστε υπόλογοι και θα πρέπει αυτά τα λίγα χρήματα που σπανίζουν να χρησιμοποιούνται σωστά και αυτό θα γίνει εφόσον οι διαδικασίες λήψης απόφασης είναι διαφανείς και στο τέλος οδηγούν σε αποφάσεις οι οποίες να λαμβάνονται συνειδητά. Οι τελικές αποφάσεις, επαναλαμβάνω, εσείς τις λαμβάνετε και εσείς έχετε την τελευταία λέξη. Αυτά αγαπητοί μου συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε μέρος σε αυτήν την προσπάθεια και που προσφέρατε τόσο στη συζήτηση. Θα παραμείνουμε σε επαφή και μέσω των κοινοβουλίων που εκπροσωπούν ε, τις, ε, τις διαδοχικές ε, προεδρίες έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι να εμπνευστούμε από την ευρωπαϊκή μας διάσταση. Ευχαριστούμε.